Okay, colleagues, we can start. You don't have to necessarily wait for more time since uh, all the key people are... Θα αρχίσουμε, συνάδελφε, λέει ο Πρόεδρος. Και ας μην έρθαν όλοι και συνεχίζουμε επομένως. Τώρα έχουμε στην μέση διάταξη το σημείο παρισμών 18 μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης. ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Τον Νοέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση τροποποίησης του σχετικού μηχανισμού για το συντονισμό και συμπλήρωση των ενεργειών των κρατών μελών όσον αφορά αυτή την πολιτική προστασία σε σχέση με τις ε, θεομηνίες που προέρχονται από άνθρωποι και εντός και εκτός της Ευρωπαϊκή Ένωσης και έτσι θα αναβαθμιστούν οι δυνατότητές μας όσον αφορά τη διαχείριση τέτοιων κρίσεων. Θα ενισχυθεί η δυνατότητα απόκρισης της Ένωσης γιατί έτσι θα υπάρχουν επιπλέον δυνατότητες για αυτό τον σκοπό σε επίπεδο Ένωσης και έτσι θα εξασφαλιστεί ότι ο μηχανισμός της Ένωσης θα είναι ευέλικτος και αποτελεσματικός. Η νομοθετική αυτή πρόταση ανατέθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος αλλά και στην Επιτροπή Περιφερειακής ε, Πολιτικής. Αλλά και εμείς συντάξαμε μία έκθεση η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και θα αφορά ε, την αντίδρασή μας σε σημαντικές θεομηνίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπάρξει επομένως συνέργεια μεταξύ πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής ενίσχυσης. Η, η της ΔΕΒΕ είναι η Ζελιάνα Ζόφκο. Έχουμε εδώ τον ε, διευθυντή της DGECO του τμήματος ε, της διαχείρισης των ε, κρίσεων, τον κύριο Γιωχάνες Λούχνερ. Έχετε 10 με 15 λεπτά. Κύριε Διευθυντά, κυρία εισηγήτρια, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος για να δώσω μια γενική έποψη των προτάσεων Να δούμε την πρώτη διαφάνεια. Με λίγα λόγια. Λέγω, με λίγα λόγια. Και τονίζω, η πρόταση αφορά την πρόληψη κυρίως. Μια που γνωρίζουμε ότι είναι ανεπαρκής στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πρόληψη όσον αφορά τις θεομηνίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και φυσικά εσείς στο μυαλό τώρα θα ανακαλέσετε τις τραγικές πυρκαγιέ των δασών του 2017, το 2016 έγινε το ίδιο, πολλά θύματα στην Πορτογαλία, αλλά έχουμε και όλε τι άλλε πλημμύρε στην Ευρώπη σε διάφορα σημεία ε, για πολλά θύματα, ανθρώπινε ζωέ, όπω και οι πυρκαγιέ των δασών. Ποιο είναι και θέμα δράση μα και εκτό συνών τη Ένωση, ε, τι γειτονιασίε, χώρε, Λοιπόν, Επομένω θα πρέπει να εξεταστείτε τι κάνουμε εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ο δεύτερο λόγο για τον οποίο υποβάλαμε αυτή την πρόταση είναι το ότι επανειλημμένο βλέπουμε δεν υπάρχει επαρκή προετοιμασία. Πυρκαγιέ, ε, επιδημίες, πλημμύρε. Δεν είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι και για την Ένωση και για τις γειτονικέ χώρες για όλα αυτά τα δίνα Και η απόδειξη είναι ότι από το 2002 ο προπολογισμό έχει εκταμεύσει πάνω από ένα δις ευρώ για αντιστάθμιση των ζημιών στα κράτη-μέλη και έχουμε φυσικά να αντιμετωπίσουμε και τους σεισμούς. Το σημερινό σύστημα βασίζεται σε έναν συνδυασμό οικονομικών πόρων. Αν χρειαστούμε παραπάνω θα πρέπει να ζητήσουμε και αν τα λάβουμε τα ελάβαμε τα παραπάνω χρήματα ή αν δεν μπορέσουμε δεν τα λάβουμε. Αν δεν τα εισπράττουμε δηλαδή θα πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι και θα πρέπει αυτή η αναμονή που σας έφερα να μειωθεί. Ε, εμείς ε, ως υπηρεσία επαγγελνούμε κάθε μέρα όλο τον χρόνο. Και αν κανείς ε, ε, θέλει να αναζητήσει αυθόρμητους δωρητές, θα πρέπει να περιμένει πολύ. Και στην Καραϊβική είχε προκύψει μια τέτοια ανάγκη και δεν μπορούσαμε να καλυφθούμε τότε για Γάλλους πολίτες. Τελικά η προσφορά υπήρξε από την Ουγγαρία, ε, για αυτό το δυστύχημα στο εργοστάσιο. Είχε προκύψει λοιπόν εκείνο το πρόβλημα στην εγκαταστάσει αφαλόντες, αλλά τελικά δεν βρέθηκε λύση αρκετά νωρί. Οπότε μιλάμε για κάποιον ο οποίο κάνει βάρδια και δύο το πρωί, θα πρέπει να κινητοποιηθεί. Και ε, δεν μπορούμε να θέλουμε να έχει και νομικέ γνώσει για να μπορεί να δει ακριβώ τι θα ισχύσει. Ε, πάντως με τη σχετική απόφαση ε, θεσπίστηκαν κάποιοι χρηματοοικονομικοί κανόνες αρκετά περίπλοκοι. Εκεί κινούμεθα, η επόμενη τώρα διαφάνεια όσον αφορά την πρόληψη και σε αυτή την αλλαγή είχαμε πάρα πολύ μεγάλες ε, τροποποίησεις και μπορείτε να δείτε εδώ στις πράσινες κουκίδες ε, τους οικονομικούς πόρους από τα διευθυντικά ταμεία που χρησιμοποιούμε για την προετοιμασία της σχετικής δράσης. Και οι μπλε κουικίδες είναι αυτά τα οποία διατίθενται από την πολιτική προστασία. Συμπέρασμα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μοχλεύσουμε, πώς θα έχουμε διαθέσιμους τέτοιους ε, πράσινους πόρους. Αυτά στην ε, ανακοίνωση διατυπώθηκαν, αλλά το θέμα είχε τεθεί και ε, με την Ρίτζο τη Γεωργία και άλλε υπηρεσίες τα λέγαμε. Θα συζητούσαμε για να δούμε πώς θα υπάρχει αυτή η κατάλληλη μόχλευση για την προπαρασκευή όσον αφορά πάντα τα διαρθωτικά ταμεία. Σε σχέση πάντα με την πρότασή μα. όταν βλέπουμε τι γίνεται διεθνώς στις ε, γειτονικέ χώρες, ε, στις χώρες της διεύρυνσης χρησιμοποιούμε το Ταμείο Πολιτικής Γειτονίας και προσπαθούμε να βελτιωθούμε αλλά όσον αφορά τις τρίτες χώρες χρησιμοποιούμε τους πόρους της ανθρωπιστικής βοήθειας ή τέλος πάντων τα κονδύλια της σχετικά με την υπηρεσία ΕΚΟ. Στην επόμενη τώρα διαφάνεια βλέπουμε για τις ε, επιχειρήσεις μας εκτός Ένωσης οπότε και θα πρέπει να λάβει την υπόψη και όσα λέει και η επόμενη διαφάνεια, αυτό το οποίο ζητούμε από τα κράτη μέλη εντό και εκτό Ένωση είναι το εξή. Να μπορούν σε αυτό το αποθεματικό, α το πούμε, ας το πούμε το εθελοντικό ε, αποθεματικό, να βάζουν τον οβολό του. Και για να είναι αυτό πιο ελκυστικό, αυξάνουμε οι διάφορε δραστηριότητε, του ρυθμού χρηματοδότηση για να διευκολυνθούν τα κράτη-μέλη να βάλουν πόρου εκεί. Και είπαμε ότι η ρυθμοί χρηματοδότησης είναι πιο αναβαθμισμένοι στα χώρες που συμμετέχουν. Όλα αυτά περιέχονται στην πρότασή μας και εκεί που υπάρχει συνεργασία για τους πόρους μεταφορών εμείς έχουμε χρηματοδότηση 100%. Πέρσι, να θυμούμε, είχαμε στην Χιλή κάποιες δασοπυρκαγιές και υπήρξε έτοιμα και στείλαμε ε, πυροσβέστες από Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία ε, πήραμε τρία αεροπλάνα, γύρισε, γύρισαν όλοι σε ένα αεροπλάνο τελικά και χρηματοδοτήσαμε 100% οπότε έτσι καλύψαμε καλύτερα το κόστος με αυτού του είδους τον κουμπαρά. Τώρα, να δούμε παρακάτω, δεν χρειάζεται να διαβάσετε όλο το κείμενο, θα σας πω, γιατί εδώ έχουμε την βασική τροποποίηση ε, του κειμένου, δηλαδή είναι το άρθρο 26, το οποίο ορίζει τα εξή. Η χρηματοοικονομική ενίσχυση για αυτές τις δράσεις, εκτός ένωσης, από τον προϋπολογισμό της πολιτικής προστασίας, δεν θα πρέπει να αποκλεί την χρηματοδότηση από άλλα εργαλεία, άλλα μέσα χρηματοδότησης της Ένωσης και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε 100% την συμπληρωματικότητα και συνέπεια αυτών των πηγών χρηματοδότησης. Τώρα, δύο πράγματα όσον αφορά το κέντρο συντονισμού. Εκεί έχουμε συγκεντρώσει όλες τις δυνατότητες αντίδρασης για την πολιτική προστασία εντός και εκτός της Ευρώπης όσον αφορά τις θεομηνίες. Και να εξασφαλίσουμε έτσι θέλουμε ότι υπάρχει αυτού του είδους η συνέπεια, η συμπληρωματικότητα. Στην πράξη αυτά Λειτουργούν πολύ καλά όπως είδαμε το καλοκαίρι στην Καραϊβική. Όπω μα είπαν οι δικοί μα, η ανθρωπιστική βοήθεια κλπ. Και υπήρξε συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφορετικών μέσων χρηματοδότηση. Παράδειγμα, στην Καραϊβική χρειάστηκε κατεπηγόντω μεταφορά και το Ολλανδικό Ναυτικό μας έδωσε ένα σκάφος, το συγχρηματοδότησε από την Πολιτική Προστασία η Ένωση και μεταφέραμε έτσι τρόφιμα από τον WF να τι πάει να πει συμπληρωματικότητα. Περί αυτού ο λόγος τώρα. Όσον αφορά το πώς θα γίνει η χρηματοδότηση της ίδιας δράσης από διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, είναι σημαντικό το θέμα του, διότι, παράδειγμα, πολλές φορές υπάρχει αίτημα για ε, φάρμακα, ιατρική βοήθεια. Έχουμε τέτοιες δυνατότητες σε διαφορετικούς βαθμούς και ευχαρίστως παρέχεται σε τρίτε χώρε αυτή η βοήθεια. Αλλά το κόστο λειτουργίας του παροχή των υπηρεσιών δεν τη χρηματοδοτούμε. Δεν μπορούμε από την κοινωνική πολιτική προστασία. Άρα, εάν υπάρχει κάποιο αίτημα και χρειάζεται τέτοια ιατρική κάλυψη, τότε τα, τα στέλνουμε, τα πληρώνουμε και συγχρηματοδοτεί η πολιτική προστασία την χώρα είναι εμπλεκόμενοι και κατόπιν έχουμε το κονδύλι ανθρωπιστικής βοήθειας ή της γειτονικής πολιτικής, ό,τι συντρέχει και αναλαμβάνει τη συνέχεια του κόστους ε, λειτουργίας. Άλλο ένα έτσι χαζούλι παράδειγμα, αλλά αυτό ήταν ε, καμπανάκι συναγερμού. Για μένα προσωπικά είχαμε ένα αίτημα από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πέρσι για ένα κινητό εργαστήριο να πάει στο Κονγκό στην, ε, σε ένα λιμάνι στην Αγκόλα, στο μέσο του πουθενά και εκεί στείλαμε έξι γερμανούς επιστήμονε από το Αμβούργο, από ένα ίδρυμα εκεί, όλα πήγανε μια χαρά. Όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει τελωνία, τα υλικοτεχνικά και ένα, και ένα από αυτά είναι το πώς θα αποχωρήσουν ε, του ιατρικού προσωπικού, ιδίως αν αντιμετωπίσουν κάποια μολυσματική νόσο και δεν προβλέψαμε όλα αυτά να γίνουν με αεροπλάνο και θέλαμε κάποιο να πάει και με το αεροπλάνο να ελέγξει, να δει τι διάδρομο προσγείωση απογείωση υπάρχει και τι μπορεί να γίνει αν χρειαστεί. Και στο Κονγκό υπάρχει συνεργασία σε αυτά τα θέματα και μου είπαν ότι δεν μπορούμε για την κένωση του προσφύγων να το χρησιμοποιήσουμε γιατί αυτό είναι πολιτική προστασία. Άρα, εν θέλουμε να εξασφαλίσουμε το ότι όπου υπάρχει προστήμενη αξία από την πολιτική προστασία να γίνει χρηματοδότηση από άλλα κονδύλια, ακριβώς για να αποφύγουμε τέτοιες δυσκολίες και για να καταστεί δυνατόν ε, οι πόροι που ξέρουμε ότι υπάρχουν και πόροι που ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να αφιερώσουν στην ανθρωπιστική βοήθεια να μπορούν να αξιοποιηθούν. Απλώς εγώ να σας πω στο ε, ε, RCC χρησιμοποιούμε την εμπειρογνωμοσύνη από αυτούς τους διαφορετικούς τομείς και θέλουμε κάποιες αρχές να γίνονται σεβαστές. Πολλά τα αιτήματα, πολλά τα αιτήματα που έχουν απορριφθεί, ας πούμε, στην Ιεμένη, είπαμε όχι στην πολιτική προστασία, ε, στο Ιράκ, σε μια πολεμική ζώνη και εκεί είπαμε όχι πολιτική προστασία, είμαστε ξαθαροί αδαμάντινοι, θέλουμε να τηρηθούν οι αρχές μας απαρέγκλητα και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, επομένως, που λέμε όχι. Εν κατακλείδη υπάρχει μια αλλαγή στο άρθρο 16 παραγράφος ένα. Αυτή η τροποποίηση αφορά μόνο την ε, διάρκεια, την προθεσμία τέλο πάντων ενεργοποίησης. Και ξέρουμε ότι σε πολλές επιχειρήσεις πρώτα-πρώτα υπάρχει το αίτημα. Τα κράτη-μέλη ω επιτοπλίστων ενεργούν τάχιστα. Όμω, αν ένα κράτο μέλο πει, Όπ, φρένο, χρειάζεται κάποιο χρόνο να τα πούμε στο Συμβούλιο, μπλα μπλα, Για ε, τότε αυτό οδηγεί σε κάτι κατάσταση. Οπότε υπάρχει αυτή η ενεργοποίηση που κρατάει έξι μήνες. Μα η πολιτική προστασία είναι κάτι που πρέπει να χρησιμοποιείται εδώ και τώρα στα κατεπήγοντα επομένω. Πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι το σύστημα θα διέπεται από κάποια νοικοκυροσύνη και δεν θα υπάρχουν κρεμότητες ε, που να κρατάνε. Άρα έτσι λοιπόν λειτουργεί αυτά το σύστημα. Κατά τα άλλα καμία ηλεκτροποίηση. Τώρα τελευταίο, μάλλον πρώτο τελευταίο slide είναι αυτό το σύνολο των εργοποίησεων το 17 ήταν 32 των κινητοποίησεων τέλο πάντων και κάθε χρόνο έχουμε διάφορες παραλλαγές συμβουλευτικές αποστολές, δασοπυρκαγιές, ε, ε, πλημμύρες, ε, τυφώνες, κυκλώνες στο εξωτερικό. Να και βλέπετε εδώ, εδώ είναι ενδιαφέρον αυτή η απεικόνηση γιατί Βλέπετε στον Άγιο Μαρτίνο τι έγινε ε, και είχαμε δύο διαφορετικά καθεστώτα νομικά που ίσχυσαν γιατί το ένα κομμάτι ήταν κοινοτική αρμοδιότητα, το άλλο όχι, αλλά τέλος πάντων καλά τα καταφέραμε και καλά τα καταφέραν και αρχές του Αγίου Μαρτίνου. Δύο. Επέμβάσεις στο Μπάνγκλα Ντες. Εκεί με την εταιρική συνεργασία συγχρηματοδοτήσαμε και μεταφέραμε επίσης και ένα κέντρο συντονισμού εκεί. Επίσης Μοσούλη στο Ιράκ. Ήταν η μεγάλη επίθεση στην Μοσούλη. Χρειαζόντουσαν φάρμακα. Δεν πήγαμε για να κάτσουμε εκεί, αλλά στείλαμε αεροπορικά τα φάρμακα. Ε, συνεργαστήκαμε με την ΕΚΟ στην περιοχή και φτάσαμε εκεί όπου ήταν ο Παγκόσμιο Οργανισμό και μετά φύγαν τα αεροπλάνα μα. Οπότε ήταν περίπλοκε και επίγουσε αυτέ οι επεμβάσει μα. Τελευταία διαφάνεια τώρα, γιατί πρόκειται για κάτι για το οποίο σίγουρα θα με ρωτήσετε και πρώτα για το ε, πόσα αιτήματα έχουμε για βοήθεια εντός και εκτός ένωσης. Ποιοι μας υποβαλούν αίτημα, βλέπετε ότι εξωτερικά ζητούν λίγο περισσότερο τη βοήθειά μας παρά εσωτερικά. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ένταση γιατί πέρσι ήταν πολύ χειρότερες δασοπυρκαγιές στην Ευρώπη από τις υπόλοιπες ε, περιπτώσεις ανάγκης. Αλλά υπάρχει βέβαια ζήτηση εκτός Ένωσης για τις υπηρεσίες μας, ιδίως όσον αφορά τους γιατρούς, μέσω του Οργανισμού Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Ε, φυσικά από χώρε που έχουν αντιμετωπίσει κάποιο είδου θεομηνία. Και ευχαριστώ. Ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε κυρία Σόφκο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λούκνερ. Ήταν εξαιρετική η παρουσίασή σας, ιδιαίτερα για την ε, μελλοντική σας δράση. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, συνάδελφοι, στην Ολομέλεια συζητήσαμε για την δράση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών που υπάρχουν όσον αφορά την αντιμετώπιση φαινομένων όπως οι πυρκαγιές ε, που πλήττουν το νότιο τμήμα της Ευρώπης. και ε, ιδιαίτερα τις περιοχές της Κροατίας, ε, της Πορτογαλίας, της Γαλλικίας. Σκοπός μας είναι να δούμε με σωστό τρόπο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων μηχανισμών και να δούμε τι αδυναμίες και τι ελλείψεις υπάρχουν. Θα ήθελα όμως να μιλήσω και για κάποιες ανησυχίες που εμπεριέχονται σε αυτή την νομοθετική πρόταση. Σας ερωτώ λοιπόν, τα κράτη-μέλη που δεν μπορούν να, να ανταποκριθούν θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση στο μέλλον, σύμφωνα με την πρότασή σας. Όσον αφορά την ανθρωπιστική αν θέλετε, πτυχή αυτών των προτάσεων. Πώς μπορούμε εμείς σαν ουδέτερος ε, ε, φορέας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, να τοποθετηθεί και να έχει μια συμπληρωματική δράση σε σχέση με όλους αυτούς που εμπλέκονται και που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Πώς μπορούμε δηλαδή εμείς σαν ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχουμε, να δραστηριοποιηθούμε, γιατί υπάρχουν χώρες όπως η δικιά μου η Κροατία που δεν μπορούν να δώσουν τις δυνάμεις τους, τα αεροσκάφη τους, χωρίς προηγουμένως να δοθεί άδεια από το Υπουργείο Άμυνας, από την πολεμική αεροπορία. Η πολιτική προστασία λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές χώρες δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική λόγω εσωτερικών προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων του συντάγματος μιας χώρας, παραδείγματος χάρη. Πρόεδρος. Η Σεσίλ και θέλει να πάρει το λόγο. Ε, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωσή σας την σημερινή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το εργαλείο για όλη την Ένωση στην Ιταλία. Από όπου προέρχομαι έχουμε πολλές θεομηνίες και πυρκαγιές. Όπως τα είπε η συνάδελφος, και έχουμε και σεισμούς και η πολιτική προστασία ανέκαθεν ναι, ήταν στο προσκήνιο κάθε χρόνο τα ίδια σε όλη τη χώρα τώρα για τις ε, πλημμύρες και για τα ποτάμια τέλος πάντων θα πρέπει και εκεί η πολιτική προστασία να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και αλλά όχι μόνο για την προστασία του κόσμου αλλά σε πολλές περιπτώσεις, όπως είπατε, θα πρέπει να υπάρχει και ο παράγων πρόληψη που είναι πολύ σημαντικός. Επομένως, αφού φτιάξαμε αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να την υποστηρίξουμε όλα τα κράτη-μέλη και να δούμε αν μπορεί να ζητηθεί από όλα τα κράτη-μέλη να κάνουν τροποποιήσεις στην εθνική τους νομοθεσία για τις θεομηνίες. Ασχολούμαι επομένως με την ε, πολιτική προστασία, η οποία ξέρω ότι έχει κάποιους περιορισμούς, κάποια όρια. Αλλά αν τα κράτη-μέλη κάνουν αυτές τις αλλαγές, τότε αυτό θα, θα πιάσει ε, τόπο, όπως τα λέει και το εγγραφό σας. Η πολιτική προστασία δεν μπορεί από μόνη της να επαρκεί, γιατί ακριβώς ε, μετράει πάρα πολύ και η πρόληψη. Άρα θα πρέπει να μην κάνουμε προς τα πίσω βήματα, θα πρέπει να βοηθούμε τις χώρες που εργάζονται όπως την ε, Ιταλία με την πολιτική προστασία. Σας ευχαριστώ πάλι και ελπίζω ότι με το έργο σας θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματική στα όσα χρειάζονται τόσα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ, η Μαρία Χόρμπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λούχνερ για την παρουσίασή σας. Η ανάλυση σας και η ανάλυση της Επιτροπής ε, συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό και βλέπουμε ότι οι μηχανισμοί που υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίνονται σε όλες τις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Υπάρχουν κράτη-μέλη που είναι πολύ πιο ενεργά, που διαθέτουν πολύ περισσότερα μέσα και σε μεγάλο βαθμό βεβαίως χρηματοδοτούν τα ίδια αυτούς τους μηχανισμούς και αυτόν τον εξοπλισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί με διάφορες πρωτοβουλίες από ό,τι άκουσα και από τις δικές σας προτάσεις να στηρίξει τη δημιουργία δυνάμεων και εξοπλισμού που να συμπληρώνουν την ε, υπάρχουσα τις υπάρχουσες δυνάμεις και εξοπλισμό στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαίως θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί και οι προτάσεις σας σίγουρα αν υλοποιηθούν θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση όλων αυτών των φαινομένων. Θα πρέπει να συμπεριφερθούμε με συνοχή, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερο συντονισμός και νομίζω ότι η πρόληψη, όπως είπατε, ιδιαίτερα για τις μεγάλες καταστροφές, είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος. Παραδείγματο χάρη στο θέμα της γεωργίας, στην επιλογή των καλλιεργειών, Βεβαίως και θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε καλύτερη οργάνωση, καλύτερη πρόληψη. Αν είμαστε λίγο πιο ε, λογική αν θέλετε στις επιλογές μας. Έχω και δύο ερωτήσεις που δεν θέλω να σας απευθύνω. Πρώτον, αυτό το RESC-EU και τα μέσα και ο εξοπλισμός εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κατάλαβα καλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δώσει το βάρος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης οτιδήποτε είναι εξωτερικές επιχειρήσεις, από ό,τι κατάλαβα θα πρέπει να γίνεται σε εθελοντική βάση. Κατάλαβα καλά. Ή και για κάποιες επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πρόβλεψη για να μπορεί να παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη ερώτηση, χρηματοδότηση. 280 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον προτείνεται. Για μένα αυτό που είναι σημαντικό είναι να πρόκειται για επιπλέον ποσά και να είναι πραγματικά επιπλέον. Να μην είναι απλώς μια διαφορετική χρησιμοποίηση ή διαφορετική ονομασία μέσων και ποσών που υπάρχουν, που ήδη θα έπρεπε να διατεθούν για αυτό το σκοπό και που ή δεν έχουν απορροφηθεί ή που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έχετε συγκεκριμένους αν θέλετε πόρους οι οποίοι θα προστεθούν στους υπάρχοντες ή από κάπου αλλού θα ανα ε, χρησιμοποιηθούν. Ε, θέλει κανένας άλλος να πάρει το λόγο? Όχι. Ε, κύριε Λούχνερ, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Για κάποιες από τις πτυχές ε, των ερωτήσεων θα ήθελα να πω ότι η πολιτική προστασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται συμπληρωματική αρμοδιότητα βάσει του άρθρου 193 και αυτό έχει συνέπειες και για τον έλεγχο και για την πρόληψη. Δεν έχουμε ούτε το δικαίωμα ούτε την αρμοδιότητα να παρέμβουμε ε, να πούμε στον κόσμο τι να κάνει, να ζητήσει εναρμόνιση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τι σημαίνει αυτό για ε, τον ε, έλεγχο και την διοίκηση των επιχειρήσεων. Δεν θέλουμε να εκχωρήσουν καμία αρμοδιότητα τα κράτη-μέλη. Το... Αυτό που παρατηρήσαμε είναι πολύ απλό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πυρκαγιές. Ο περίοδοι όπου υπάρχουν κίνδυνοι πυρκαγιών. Έχουμε επαρκείς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, ε, στην Ιταλία. Το θέμα είναι ότι αν όλε αυτές οι χώρες ε, πλήττονται ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο την ίδια περίοδο από μια, φυσική, από μια συγγνώμη, ε, πυρκαγιά δάσους, ε, τότε δεν μπορεί κανείς ε, ως εθνικός πολιτικός να στείλει ένα αεροσκάφο στο παρελθόν ε, ακόμη και τον χρειάζεται στη χώρα του επειδή ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος οπότε το σημαντικό είναι να υπάρχουν πόροι που είναι διαθέσιμοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι υποχρεωτικά ένα στόλο, αλλά κάποιο είδου τέλο πάντων πόροι που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μία άλλη λύση είναι να το καταστήσουμε πιο θελκτικό, να συγκεντρώνουμε περισσότερου πόρου ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και θέλω να τονίσω ότι αν ένα πόρο βρίσκεται σε αυτό το καλάθι πόρων και κάποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που χρειάζεται για εθνική ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, ένα πόρο, τον κρατά στο, στη χώρα του και το χρησιμοποιεί. Δεν ζητούμε δηλαδή να ε, έρθουμε εμείς και να ελέγξουμε οποιοδήποτε τρόπο ε, διαχείρισης των πόρων, ούτε σας ζητούμε συντονισμό σε εθνικό επίπεδο. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει μία εφεδρική ικανότητα που να δημιουργείται. Εμεί θα λάβουμε την απόφαση μόνο κατόπιν ε, αιτήματο των κράτου μέλου, όχι μονομερό και βέβαια ε, επιχειρησιακό έλεγχο έχει η χώρα η ίδια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να μπούμε στα χωράφια των εθνικών επιχειρήσεων καθόλου, ούτε ζητούμε να, έχουμε, να, να βάλουμε πόδι τέλος πάντων στους εθνικούς πόρους. Όσον αφορά τώρα την ανθρωπιστική βοήθεια και το τι κάνουμε σε σχέση με μάλλον από κοινού με του, τις υπηρεσίες του ΟΗΕ ε, που μας ζητούν βοήθεια όπως ο ΠΟΗ για παράδειγμα, ε, τη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού. Ε, αυτή είναι βασική μας εταίρη. Τι κάνουμε διαπραγματευόμαστε κάποιες τυποποιημένες διαδικασίες επιχειρήσεων εγώ έχω μάλιστα και παρελθόν στην ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχει μια ανάμιξη πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ε, είναι συνεργάτες μας, ε, οπότε... Εντάξει, είναι κάπως ε, στο αίμα μας κατά κάποιο τρόπο το κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά Υπάρχουν επίγουσες καταστάσεις πάρα πολύ περίπλοκες ε, και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν άνθρωποι πολιτικής προστασίας που εμφανίζονται με κάποια στολή και δεν μπορεί να πάει κανείς ας πούμε ε, σε μια εμπόλεμη ζώνη αλλά ε, στις συμφωνίες μας με τους διεθνείς οργανισμούς μπορούμε να συμπεριλάβουμε πότε θα χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι πολιτικής προστασίας. Προς την Ιταλίδα Ευρωβουλευτή, το είπα στην αρχή, είναι εν μέρη ζήτημα χρηματοδότηση, γιατί ε, το μεγαλύτερο τμήμα τη χρηματοδότηση προέρχεται από το διαρθρωτικά ταμεία. Υπάρχει όμω και το ζήτημα τη αρμοδιότητα, που είναι το βασικότερο. Μπορούμε έτσι να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την πρόληψη και την ετοιμότητα και, τι σχετικέ και τις σχετικές δαπάνες. Ενθαρρύνουμε σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και κάποια αιρεσιμότητα. Ε, θέλουμε να το βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι και αυτό θα είναι τμήμα τη πρόταση για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο που θα υποβάλει την Άνοιξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πρόταση τη δική μας, αυτή η αυτή, επειδή είναι μια συμπληρωματική αρμοδιότητα, αυτό που ζητούμε εμείς, ε, ζητούμε γενικές εκθέσεις για τα σχέδια ετοιμότητας των κρατών μελών για τα σχέδια πρόληψης και θα έχετε διαπιστώσει ότι υπό την τρέχουσα νομοθεσία ως προς τα ε, σχέδια διαχείρισης πρέπει να τα έχουν τα κρατη αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να τα στείλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι απλώς να τα ζητούμε. Αν δούμε ότι ένα κράτος μέλος ε, χρόνο με το χρόνο αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, τότε έχουμε εισαγάγει μία διάταξη η οποία λέει ότι σε αυτή την περίπτωση αφήστε μας να ρίξουμε μία ματιά στα σχέδια διαχείρισης και ετοιμότητά σας και να κάνουμε και ένα διάλογο. Για το ερώτημα τώρα της Γερμανίδας ε, Ευρωβουλευτού. Το ζήτημα της διάσωσης είναι σημαντικό. Το να υπάρχει λοιπόν μια εφεδρική ικανότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λογικό. Η λογική τώρα για το κομμάτι που αφορά το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διτή. Πρώτον, αύξηση των πόρων, στο καλάθι των πόρων, ε, θα υπήρχαν ε, και κάποια οικονομικά κίνητρα γι' αυτό, αν εγκριθεί ε, η ε, συμφωνία και δεύτερον χρήση άλλων δημοσιονομικών γραμμών και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα των κρατών μελών ε, είτε θα είναι η ανθρωπιστική γραμμή του προπολογισμού είτε οποιαδήποτε άλλη που θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό. Το πρόβλημά μας για την ώρα είναι ότι νομικά φαίνεται δύσκολη ανάμειξη των δύο. Για το κομμάτι που αφορά το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε να έχουμε αυθόρμητες προσφορές ε, μάλλον δεν θέλουμε αυθόρμητες προσφορές, θέλουμε να υπάρχει ένα καλάθι πόρων που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να μην έχουμε το πρόβλημα που εμφανίστηκε το καλοκαίρι ότι έχουμε πόρους αλλά δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτούς ε, άμεσα οπότε οι ενδιαφερόμενες χώρες ε, ε, στρέφονται αλλού και παίρνουν συγχρηματοδότηση από άλλες γραμμές προϋπολογισμού. Να σας πω την αλήθεια όλα αυτά συζητώνται και στο Συμβούλιο, αλλά εξ όσων γνωρίζω και όσον αφορά τα αεροσκάφη ε, για τις πυρκαγιές. Ε, οικονομικά το συζητήσαμε το θέμα αυτό και πέρσι, το εξετάσαμε. Δεν είχε νόημα να πάμε στη χιλία, ας πούμε πέρσι για τα 290 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, ναι, 260 προέρχονται από το μέσο ευελιξίας, όχι από άλλες γραμμές προπολογισμού περίπου 260 εκατομμύρια και περίπου 20 εκατομμύρια από άλλα προγράμματα, αλλά ναι. όχι από τον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Είναι κάποια υπόλοιπα, μικρότερα. Όμως το μεγαλύτερο τμήμα προέρχεται από το μέσο ευελιξίας. Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός, μετράω τα λόγια μου, είναι φρέσκο χρήμα, αλλά υπό το τρέχον πι δελτα πι. Οπότε δεν ε, είχαν ε, ε, δοθεί αυτά τα χρήματα στο παρελθόν. Υπάρχουν όμως υπό το συγκεκριμένο, υπό το τρέχον πι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Τσοφκό έχει τον λόγο να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατα... Εξηγήσατε νομίζω πολύ καλά ποιες είναι οι προθέσεις. βεβαίως θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. ευχαρίστως να μιλήσουμε και διμερός ε, να ε, καταλάβω καλύτερα τι ακριβώς είναι αυτή η συγκέντρωση των πόρων. Αυτό σημαίνει ότι χάνουμε ως προς την ικανότητα ε, και ως προς την ενίσχυση το, της πολιτικής προστασίας εντός της χώρας μας, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε ένα, πλεονό, να έχουμε ένα μειονέκτημα ε, για τη δική μας πολιτική προστασία που μπορεί να συμβαίνει αν δημιουργήσουμε αυτήν την εθελοντική συγκέντρωση πόρων και αγοράζουμε και νέους πόρους. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Δεν θα θέλαμε πάντως να συμβεί κάτι τέτοιο. have to ask... Και τώρα να κάνω μία ερώτηση. Ο κύριος Στάινερ είναι εδώ. Α, ναι. Είστε εδώ. Δεν είστε. Yeah, colleagues, uh... Συνάδελφοι, θα αργήσει ο προσκεκλημένος μας. Άξο θα είναι εδώ παρά 20 και 4 παρά 20. Θα κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα. σε ευχαριστώ.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 Um, so I don't know what's happened because Ms Stein has left the EAS now, so it's not very far. So Υπομονή γιατί ε, είχαν πάει προσκεκλημένοι μας στην Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης που είναι λίγο πιο πάνω. Είναι λίγο μακριούτσικα, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε τόσο πολύ. Μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα και βλέπουμε.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

AUTHORWAVE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

Okay, colleagues, we can now resume our committee. Um, moving... Συνεχίζουμε συνάδελφοι και προχωρούμε στο θέμα 19, το οποίο είναι συζήτηση με τον Αχίμ Στάινερ. Είναι ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Αχίμ Στάινερ. Ε, ήταν στο Συμβούλιο, το άτυπο Συμβούλιο για την ανάπτυξη, άργησε και εμείς αργήσαμε, η μία καθυστέρηση έφερε την άλλη και, το γεύμα εργασίας καθυστέρησε, ε, επομένως ε, ήρθε αργά και θα πρέπει τώρα να καλύψουν το χαμένο χρόνο για τη δική μας συζήτηση. Με χαρά μας σας αντίσαμε στην Υόρκη και εσείς ήσασταν πολύ φιλόξενος σε εκείνο το φόρουμ ψηλού επίπεδου. Και τώρα έχετε στο χαρτοφυλάκιό σα και τους στόχου στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη και ένα σωρό άλλα θέματα και τα είπατε με τους υπουργού, πάντως και πάλι καλώς ορίσατε ε, και καλώς και οι προσκεκλημένοι μας οι βουλευτές από την Γκάμπια είναι από διάφορες επιτροπές ε, και ανεδείχθησαν από τις πρώτες ελεύθερες εκλογές της χώρας, τις πρώτες 25 χρόνια, να, και μερικά καλά μαντάτα. Μας χρειάζεται μια τέτοια φρέσκια δημοκρατία που φέρνει την ελπίδα μαζί της θα ζητήσουμε τώρα για αυτούς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και θα ακούσουμε και τον κύριο Μούσα Μουλιάση, τον επικεφαλή σας, αργότερα για να μας εξηγήσει τα της νεαρής δημοκρατίας σας και για τα των SDG, των στόχων αυτών της ανάπτυξης, αλλά η σκητάλη πρώτα στον κύριο Στάινερ. Ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα, πρόεδρε. Ευχαριστώ εσάς και συγγνώμη από όλους σας που άργησα. Αυτό είναι κάτι επικίνδυνο να το κάνει στο κοινοβούλιο. Αλλά ξέρετε τα κράτη-μέλη σας με κλειδώσανε στην αίθουσα και απόδραση δεν ήταν δυνατή. Αλλά ελπίζω ότι θα αποσμηθώ από τις συζητήσεις. Και θα συνεχίσουμε σήμερα την συζήτησή μας που βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που την κάνουμε ούτε θα είναι η τελευταία και ήρθα να τα πούμε για να δούμε πώς θα αναβαθμίσουμε αυτή την εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοινοβουλίου, Κομισιών και του ΟΗΕ γιατί είναι ταραγμένη η καιρή που ζούμε είναι καιρή αποσταθεροποίησης, ανησυχίας γιατί έχουμε πολλούς παράγοντες ε, αστάθειας πολλούς παράγοντες που οδηγούν σε σύγκρουση, προστριβή Βέβαια έχουμε και ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είδαμε στο τη Αφρικής και όλα αυτά προβληματίζουν και ανησυχούν. Δεν είναι θέμα απεσιόδοξης οπτικής για τον κόσμο, αλλά όπως και ο Γενικός Γραμματέα, όπως και εσείς, όλοι γνωρίζουμε ότι η τελευταία διετία, αλλά και η προοπτική για την επόμενη διετία, αφορούν μια συγκυρία που με τίποτα δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Δεν είναι, α, τον έχει κάποια προστριβή εδώ, ένα, μια άλλη μικρή σύγκρουση εκεί, αλλά πρόκειται για κάποιο είδους ε, διάβρωση των βασικών αρχών. Και πάντοτε υπάρχουν διαφορές ε, απόψεων, αλλά μιλούμε τώρα για υπονόμευση των αρχών που είναι η βάση της συνεργασίας μας. Είναι το θεμέλιο θεσμικών οργάνων όπως ο ΙΕ, η Γενική Συνέλευση, η και το Συμβούλιο των ε, Δικαιωμάτων. Επομένως έχει διαταραχθεί η αίσθηση της τάξης που διέπει τον κόσμο και που αφορά όλες τις δυνάμεις που συνθέτουν αυτόν τον κόσμο και σε πάρα πολλές χώρες ε, ο κόσμος σε αυτές τις αρχές στηριζόταν. Αν κανείς μια ματιά στον έξω κόσμο θα διαπιστώσει πρώτα πρώτα τον αγώνα που δίνει η Ευρώπη για να μείνει στην επιφάνεια. Μετά πάμε προς τον νότο και βλέπουμε μια περιοχή που σήμερα μαστίζεται από εντάσεις, από συγκρούσεις, από εμφύλιες προστριβές, χωρίς προηγούμενο. είδαμε ποιες είναι οι συνέπειες της συγκρούσης στην Συρία, αλλά δεν είναι μόνο εκεί το θέμα είναι σαν ο μισός κόσμος εναντίον του άλλου μισού. Και είχα πάει στο Κουβέιτ, συζητήσαμε και για το Ιράκ, την ανασυγκρότησή του, να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα αναχαιτήσουμε το Ισλαμικό κράτος, πώς η περιοχή θα επανέλθει στην ομαλότητα και τώρα είπαμε ότι πάμε για 88 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι το κόστος αυτής της ανασυγκρότησης. 40 από τις απελευθερωμένες πόλεις ισοπεδώθηκαν από βομβαρδισμούς, από τις μάχες γενικότερα. Και για να γυρίσει ο κόσμος σε αυτές θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες προς τούτο. Ήμουνα δύο μέρες στην Βηρητό. Είδα μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται επίσης από ευαισθησία, είναι πολύ ευάλωτη και κατά κεφαλή έχουν τους περισσότερους πρόσφυγες. Η Ένωση όπως και ο ΙΕ βοηθά τον Λίβανο για να φέρει το βάρος των παραπάνω προσφύγων πέραν των Παλαιστινίων. Όλα αυτά είναι κατεπίδοντα, είναι πιεστικά. Τις τελευταίες δύο μέρες αυτά κουβεντιάζουμε εδώ στις Βεξέλλες διότι αλλιώς η θέληση, η δυνατότητα για να συγχυστεί η φιλοξενία του Λιβάνου για να μπορέσει να αποτελεί ο λοιπόν καταφύγιο με την πραγματική έννοια ε, δεν μπορεί να είναι κάτι που δεν αλλοιώνεται λόγω των συνθήκων. Όλα αυτά σας τα λέω προσαγωγικά για τους στρατηγικούς στόχους, για τη βασική τάση αυτών των στόχων και τη θυματολογία του 2030 βασίζεται στη διασύνδεση των μεταβλητών των διαφόρων θεμάτων, να καταλάβουμε ποια είναι η πηγή των συγκρούσεων, του ριζοσπασ... της ριζοσπαστικοποίησης, γιατί όλα αυτά είναι μέσα στην κοινωνία μας. Και δεν μιλούμε εδώ μόνο για χώρες μέσα Ανατολής και Βορείου Αφρικής. Περιθωριοποίηση, ριζοσπαστικοποίηση, εξτρεμισμός. Εδώ, στην καρδιά της Ευρώπης η αποξένωση των νέων. όλα αυτά που το εισπράττουν ως ένα σύστημα που έχει χάσει την αξιοπιστία. Δεν μπορούν φανταστούν πώς θα πάει η ζωή τους. Μέσα στην ανεργία, μέσα σε μια πολιτιστική μειονότητα. Ε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ δηλητηριώδη και διαβρωτικά. Οπότε έτσι αναδύονται αυτοί οι στόχοι της ανάπτυξης αυτό προέκυψε το 2015 ή το καλοκαίρι του 12 αν θέλετε. Ε, αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό αναδύθηκε μέσα από την κρίση, μέσα από την αραβική άνοιξη, από το ότι όλο ένα και περισσότεροι συνειδητοποίησαν ότι η μη βιωσιμότητα και η ανισότητα άρχισαν να γίνονται κάτι το μόνιμο στον αγώνα για οικονομική πρόοδο, για όλη την κοινωνία. Το 2015 τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ ψήφισαν για αυτό το θέμα το 2030. Όμως τότε δεν ξέρανε ότι θα υπήρχαν και αντίρροπες δυνάμεις. Χρειάζεται αύξηση του ΑΕΠ, χρειάζεται απορρίθμιση των αγορών να, για να πετύχει η παγκοσμιοποίηση που θεωρητικά έπρεπε να οδηγήσει στην οικονομική επιτυχία, το κόστος των επιπτώσεων ε, στο περιβάλλον, το τίμημα για να προχωρήσουμε, για να επαναπροσδιορίσουμε το μέλλον μας. Οπότε, είπαμε ότι ε, το 2000 άλλαξαν πάρα πολλά και σήμερα βλέπουμε ότι ο κόσμος διψά για να ξαναέχει ελευθερία επιλογής. Οικονομία και κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον αυτά θα πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Θα έπρεπε αυτά να είναι, να είναι το περιεχόμενο της εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα. Ιδάλλως έχουμε αποξένωση από αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς πρώτα-πρώτα. Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, ένωσης ΟΙΕ, είναι πάρα πολύ κρίσιμες στιγμές η Ένωση είναι ένα πείραμα. Τι πάει να πει πολυμέρεια. Στο επίκεντρο είναι η ενότητα, η πολυμορφία και όλα τα άλλα μετά που ανεβήθηκαν όπως η επικουρικότητα, η συμπληρωματικότητα. Τελικά είναι όμως ένα πείραμα. Το δηλαδή μαζί καταφέρνουμε περισσότερα από όσα ο καθένας μόνος του. Ο ΙΕ είναι μια ευρύτερη, μεγαλύτερη εκδοχή τούτου μεγαλύτερη διαφορετικότητα, μεγαλύτερες παιδικές διαφορές και περισσότερες ανισότητες. Οπότε έχουμε τώρα αυτή την ε, διοίκηση που έχει πολλές επιφυλάξεις στην Αμερική. Έχει πολλές επιφυλάξεις για την ε, διεθνή κοινότητα. Επίσης σήμερα η σχέση μεταξύ του που δεν τα πήγε καλά η ανάπτυξη αλλά και οι συγκρούσεις που ξεκινούν και ο εξτρεμισμός, όλα αυτά έχουν συνδεθεί περισσότερο από ποτέ. Οπότε απευθυνόμενος σε εσά θέλω να κάτσετε και να αναθεωρήσετε τους στόχους SDG. Θα πρέπει να καλυφθούν οι κορυφαίες μας προτεραιότητες για την ανάπτυξη. Αυτό είναι πρώτα-πρώτα πλαίσιο για την ανάπτυξη. Για μια ανάπτυξη που πάει παραπέρα από την οικονομική ανάπτυξη κοινωνική ισότητα, περιβάλλον, βιωσιμότητα, να πάμε και προς αυτές τις πτυχές. Αλλά και η παγκοσμιότητα. Αυτό πάνε να πει η SDGs. Δεν είναι μόνο θέμα το τι γίνεται στην Κάμπη, είναι και το τι γίνεται στη Γερμανία, στην Κίνα, στη ΣΥΠΑ. Έχουμε αυτούς τους παγκόσμιους στόχους που έχουν σχέση με θεμελιώδεις αρχές, ούτως ώστε να πετύχει αυτή η ανάπτυξη να βελτιωθούν οι ιδιωτικές συνθήκε, η παιδεία, οι υποδομές, επίσης και η κοινωνική συνοχή. Εάν δεν κανείς τίποτα για την ανισότητα σε μια κοινωνία, τότε θα ανατραπεί αυτή η, κοινωνία, θα υπονομευθεί. Πήγα σε Αιθιοπία, πήγα σε Σομαλία και μιλήσαμε για την αλλαγή του κλίματος είδαμε τα ακραία φαινόμενα όπως οι ξηρασίες. Αυτά δεν είναι μόνο θεωρητικά. Το κύριο Αφρική Αφρικής και η Αιθιοπία τώρα έχουν περάσει μια μακρά περίοδο ξηρασίας που είναι πολύ χειρότερη από ότι τη δεκαετία του 80 ακριβώς γιατί μαζί προσπαθήσαμε να δούμε τι διαχείριση θα κάνουμε για τις θεομηνίες επειδή με την Κομισιόν και με τον ΟΗΕ κινητοποιηθήκαμε από πέρσι έχουμε αυτό το εργαλείο της αντίδρασης και μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τους λοιμούς πέρσι. Οπότε έτσι έχουμε το θεματολόγιο της ανάπτυξης για μια τέτοια αντίδραση στα κάτι επίγοντα αλλά και με μακρόπνο χαρακτήρα σαν στρατηγική. Και οπότε έτσι και στον ΟΗΕ το πρόγραμμά μας για την ανάπτυξη έχει ένα στρατηγικό πλάνο ούτως ώστε τα SDG να είναι το θεμέλιο για την επόμενη γενιά τέτοιων ε, προγραμμάτων και για το σύστημά μας που έχουμε. Πάνω από 104 χώρες έχουν ζητήσει να καλυφθούν από ένα τέτοιο σύστημα, δηλαδή να αναδεχτούν σε εθνικό επίπεδο και στο τοπικό επίπεδο αυτούς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στα γραφεία του Πρωθυπουργού έχουν και γραφεία ανάπτυξης για αυτούς τους στόχους. Αναζητούνται ε, συμμαχίες, ε, συνεργασίες ε, μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και δήμων, ούτω ώστε να αναλυθεί δράση σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, αναζητούμε αυτούς τους στόχους σαν πλαίσιο για κινητοποίηση πόρων πέραν των δημοσιονομικών και για όλες τις χώρες. Να μην ξεχνούμε ότι ο δημόσιος κορβανάς είναι λιγότερο του 20% των δαπανών στην οικονομία. Και αν θέλουμε να πετύχουμε για αυτό το μετασχηματισμό και να πάμε σε οικονομία με λίγο άνθρακα, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε σε επόμενη ετία όλες τις ευκαιρίες για την Αφρική και άρα χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, των ε, εθνικών χρηματοοικονομικών αγορών και πόρων. Ε, όλα αυτά είναι απαραίτητα. Ίσως έχετε ακούσει αυτά από την Οικονομική Επιτροπή Αφρικής, όπου τα αποθεματικά είναι χίλια δις τώρα και 600 από αυτά τα δις δεν, ε, ε, δεν επενδύονται εκεί. Αυτά τα 600 δις πάνε στα χρηματιστήρια. Νέα Υόρκη, Ζηρίχη, Χονγκ Ε, αυτό δείχνει την πρόκληση των διαθέσιμων αποθεματικών και τη δυσκολία με τις επενδύσεις. Άρα, έχουν πολλή δουλειά μπροστά μας για να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα. Και θεωρούμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε τις κυβερνήσεις για να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις σε κάποιες χώρες έχουμε κάποια εργαστήρια καινοτομία για τους στόχους SDG. Έτσι το λέμε και μπορούμε να συγκεράσουμε τη δράση Υπουργείων, ιδιωτικού τομέα, τις ιδέες τους, την δημιουργικότητα, think tank, πανεπιστήμια, πανεπιστημιακών και έτσι επιταχύνεται η υλοποίηση των νέων προσεγγίσεων. Και αυτό για ποιο λόγο είναι σημαντικό, διότι οι στόχοι έχουν θεμέλιο κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Το ότι αν επενδύσει κανείς σε έναν στόχο, θα πρέπει τότε να υπάρχει απόδοση και επίδοση και σε άλλο στόχο. Άρα, θα πρέπει και η οικονομική πολιτική να είναι συμβατή με τους στόχους μας. Να πιάνει η ομορφιά του πλαισίου των στρατηγικών στόχων. Γιατί έτσι είναι πιο ξεκάθαρο το ότι όταν μιλούμε για μείωση του άνθρακα στην οικονομία, αυτό μας οδηγεί σε μια πιο καθαρή ενέργεια, Φερρυπίν, για την Αφρική. Και στο ότι στρεφόμαστε έτσι στις ανέβνες πηγές ενέργειας και βοήθειας έτσι προς την Ήπεθρο, όπου ζουν οι περισσότεροι στην Αφρική. Έτσι δίνουμε επομένως πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης και έτσι με μία επένδυση κανείς καλύπτει τους τέσσερις στόχους. Να η διαφορά σε σχέση με το κλασικό αναπτυξιακό μοντέλο. Και έτσι μπορούμε να διαχειριστούμε τους πόρους. πόσο αυτά θα πιάσουν τόπο στην κοινωνία των πολιτών, στον ιδιωτικό τομέα κλπ. Οπότε, με το δικό μας πρόγραμμα εκφράζουμε τον ρόλο μας, όπως το βλέπουμε, ότι να μην εστιαζόμαστε μόνο στις χώρες που περνάνε κρίση και είναι λιγότερο ανεπτυγμένες αποτελούν πλαίσιο αυτή στόχη για κάθε χώρα. Άρα, το ίδιο σημαντική είναι η δουλειά μας και στις χώρες μέσω εισοδήματο. Το ίδιο σημαντική όσο και στις χώρες που είναι πιο φτωχές. Γιατί οι περισσότεροι φτωχοί ζουν στις χώρες με μεσαίο εισόδημα. Και οι περισσότερες κρίσεις που έχουμε σήμερα προέρχονται από μη βιωσιμότητα, από ανισότητα, από κακή διακυβέρνηση, από τις χώρες μεσαίου εισοδήματος. Ε, επομένως, το κριτήριο του κατακεφαλήν ΑΕΠ αυτό δεν θα ήταν ο πιο δόκιμος τρόπος για να δούμε το θέμα. Φυσικά και υπάρχει σπάνιση στους πόρους, θα πρέπει να κάνουμε επιλογές, αλλά πολύ συχνά οι σημερινές μας επιλογές λαμβάνουν υπόψη της ε, αποτυχίας μας σαν κάτι που προκύπτει έτσι μαγικά. Θα πρέπει κανείς να δει του ευρύτερου τοπίου, δηλαδή από πού πηγάζει ο εξτρεμισμό. Εδώ και δεκαετίες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και ακραίε συνθήκε και για αντίδραση στα κατεπήγοντα. όμω ταυτόχρονα χρειάζεται να δούμε τι θα κάνουμε με την ριζοσπαστικοποίηση. Οπότε σήμερα περισσότερο από την τελευταία 30 ετία ξέρουμε πολύ περισσότερο, 100 φορέ περισσότερο για μια ειρηνευτική δύναμη για ανασυγκρότηση, για ανάπτυξη δυνατοτήτων, θεσμών κλπ. Οπότε ανάπτυξη, ειρήνη και σταθερότητα, όλα αυτά είναι διαφορετικές πηγές αλλά αλληλένδετες. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι οι στόχοι SDG είναι το κατάλληλο πλαίσιο. Ούτως ώστε να μην έχουμε όρια διοικητικά, γραφειοκρατικά, για να μπορούμε να προχωρήσουμε το έργο μας. Χρειάζεται επομένω για την ανάπτυξη, επενδυτική πολιτική, με ούτω ή προληπτικό χαρακτήρα. Και αυτό ακριβώς είναι το όραμα του Γενικού Γραμματεία Κουτέρες για το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν όμως και λύσεις. Και αυτό είναι το μήνυμα. Ήμασταν ε, με δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες ε, στην Αφρική, η μία στη Σενεγάλη, η άλλη στην ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και συναντήσαμε και τις αποστολές για τη διατήρηση της ειρήνης. Η προσπάθεια αυτών που συναντήσαμε να συνεισφέρουν στην προσπάθεια εκδημοκρατισμού των χωρών τους και φυσικά στην ανάπτυξη και αυτό το μήνυμα που όλοι μας είπαν είναι ότι χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση ανάπτυξη. Οι προοπτικές λοιπόν είναι κάτι που φυσικά και μας απασχολούν, αλλά δεν ξεχνάμε ότι χρειάζεται συνεργασία και με τις δυνάμεις αυτές ασφαλείας. Θα ξεκινήσουμε τώρα με το των ομιλητών. Ναι, συναντηθήκαμε και στην ε, Νέα Υόρκη. Ήταν μαζί και ο κύριος Βέντα. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω γιατί θεωρώ ότι πραγματικά εμείς ε, σαν ε, μέλη του Κοινοβουλίου θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και για αυτά που μας είπατε, αλλά γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι με αυτή την ταινία μπορούμε να δούμε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο αυτό το θέμα. Η πολιτική της ανάπτυξης ε, έχει όρια τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε. Και αυτό μας καλείται να κάνουμε. Παραδείγματο χάρη, ξέρουμε ότι θέματα που αφορούν το εμπόριο, που αφορούν την κλωστοεφαντουργία, Παραδείγματο χάρη, και οι στόχοι, η αναπτυξιακοί, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να μπορέσουμε και σε τομείς όπως παραδείγματος χάνει κλωστοεφαντουργία, να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις αδυναμίες, να συνδυαστούμε παραδείγματο χάρη με τα Ηνωμένα Έθνη, να περάσουμε από τομείς τόσο διαφορετικούς όσο είναι παραδείγματος χάρη το περιβάλλον, οι εμπορικές σχέσεις και φυσικά να μάθουμε ημέν από τους δε. Σε αυτήν την διακοινοβουλευτική συνεδρίαση που είχαμε με μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων της Αφρικής θα θέλαμε να ξέρουμε αν έχετε τέτοιου είδους εμπειρίες, πώς δηλαδή μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα με τα Εθνικά Κοινοβούλια και πώς εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει, να συνεισφέρει, Έχουμε μια εμπειρία με την Καραϊβική, έχουμε μια εμπειρία με την ε, Λατινική Αμερική, όπου έχουμε σε αυτά τα πλαίσια συνεργασία, αλλά εσείς τι μπορείτε να μας πείτε, γιατί πιστεύω ότι σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναπτύξουμε τέσσερις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες και αλλού. Έχουμε και την Μπάρμπαρα, η οποία είναι πολύ καλή αν θέλετε, όσον αφορά τη συνεργασία με την Επιτροπή μας, φίλοι της Επιτροπής, δεν είναι η πρώτη φορά που έχετε εδώ και πριν την επόμενη συνάντηση κορυφής του Πολιτικό Φόρουμ, είναι πολύ σημαντικό να συσφίξουμε τους δεσμούς μας, να βελτιώσουμε την συνεργασία. Γι' αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που Ζωζε Φάρια είναι εδώ, είναι σκιώδης της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος για τα θέματα των ε, στόχων και με μεγάλη χαρά τον καλωσορίζουμε σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι οι δύο μας επιτροπές θα πρέπει να συνεργαστούν ε, περισσότερο και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Στα πορτογαλικά είχα προβλέψει να σας τα πω, αλλά σήμερα δεν προβλέπονται τα πορτογαλικά στο καθετό διερμηνίας. Μπορεί λοιπόν να κάνω κάποια λάθη. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Ελπίζω να είστε ποιητικοί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Στάινερ ε, για την παρουσία του, όπως επίσης και για την, τον σημαντικό και πολύ ενθαρρυντικό λόγο σας, την πολύ ενθαρρυντική ομιλία σας. Ξέρετε ότι είμαι Πορτογάλος ε, Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ ε, και είμαι ε, τακτικό μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ε, θα επικεντρωθώ λοιπόν περισσότερο στο περιβάλλον. Ήμουν η συγητής ε, της έκθεσης της Διεθνούς Διαχείρισης των Ωκεανών βάσει των στόχων του 2030. Ήμουν και στη Νέα Υόρκη για τη διάσκεψη για τους ωκεανούς. Ήμουν επικεφαλή αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαι και σκιώδη εισηγητής ε, της έκθεση της Ευρωπαϊκή Ένωση για ε, την ε, αηφορία. Θέλουμε να δείξουμε ιδιαίτερα τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πλήρωση των ε, στόχων του 2030 στο πλαίσιο του, ε, ε, των στόχων αηφόρου ανάπτυξης είναι γεγονός ότι η περιβαλλοντική και κλιματική διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτύξει έναν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του θεματολογίου για το 2030 στην προσπάθεια εξάλληψης της φτώχειας, όχι μόνο στο πλαίσιο των 17 στόχων, αλλά και στους υπόλοιπους 169 συνδεδεμένους στόχους που καλύπτουν κάθε πτυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους Συμφωνίας των Παρισίων εισηγητής για την έκθεση της δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αηφορία που μας δίνει μια μοναδική δυνατότητα να τοποθετηθούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, ευρωπαϊκή δράση δηλαδή για την αηφορία. Και Βέβαια, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει κάποιες, κάποιοι συμβιβασμοί σε σχέση με το ψήφισμα της 16ης Ιουλίου του 2017, ε, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Ε, έχουμε καθορίσει έναν ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο για τους στόχους της αηφορίας ε, και ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2030 αποτελεσματικής και πλήρους ε, παρακολούθησης, ε, συστήματος παρακολούθησης και εφαρμογής των αναπτυξιακών στόχων αηφορίας για το 2030. Γι' αυτό ακριβώς εμείς ζητήσαμε από, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σεβαστεί ε, τις, ε, ε, το θεματολόγιο αυτό, όπως επίσης και το σχέδιο εφαρμογής του Βουσκού του 2002, όπως επίσης και των συστάσεων της διάσκεψης του ΟΗΕ για το θεματολόγιο των αναπτυξιακών στόχων αηφορίας μέχρι το 2030. Οι εξωτερικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα έπρεπε να είναι συμβατές ε, με τους στόχους αηφόρου ανάπτυξης ε, και ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι εξωτερικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους στόχους αηφόρου ανάπτυξης ε, και δεν αντιβαίνουν στην ανάπτυξη κάποιων περιφερειών όπως για παράδειγμα των υποανάπτυξη χωρών. Σας υπενθυμίζω το ψήφισμα του 2017 και πάλι που κάλεσε επιγόντω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μία πρόταση για μία διαδικασία που συμπεριλαμβάνει τη διαδικασία νομοθεσία την αναθεώρηση της, να υπάρξει ένα περιεκτικό μια περιεκτική στρατηγική ανάπτυξης ε, και βέβαια η πρόταση που ενεκρίθη στις 6 Ιουλίου ήταν πάρα πολύ φιλόδοξη. Ε, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην κλιματική αλλαγή και στην ε, απαλυφή του άνθρακα από την οικονομία, στην κυκλική οικονομία και την αποδοτικότητα των πόρων, την προώθηση της καινοτομία της επιστήμης και τεχνολογίας, ε, την διατήρηση των φυσικών πόρων και την ολοκλήρωση το, του θεματολογίου των ευρωπαϊκών εξαμήνων, την αντιμετώπιση των ανισο, τον εντός και μεταξύ των κρατών μελών και την ενσωμάτωση ε, των πιο περιθωριοποιημένων και των πιο μειονεκτούντων. Όλα αυτά τα είπατε, όμως δεν είναι αυτά αρκετά κύριε Στάινερ. Ε, ε προφανώς θέλουμε αυτοί οι στόχοι να συμπεριληφθούν σε μια ευρύτερη προσέγγιση που θα έχουμε, όμως η συνεισφορά ε, των εμπλεκομένων φορέων, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι απαραίτητη. Η παγκόσμια δράση είναι απαραίτητη γιατί ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο και τώρα περισσότερο από ποτέ βλέπουμε ότι κάποιες χώρες απομακρύνονται σε σχέση με τους στόχους αυτούς όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε για παράδειγμα. Έχουμε μεγάλες αμφιβολίες μπροστά μας σε σχέση με την πραγματική ικανότητα του ΟΗΕ να επιτύχει τους στόχους ε, του 2030. Ε, αναφερθήκατε στον κύριο Γκουτιέρε που είναι συμπατριώτης μου. Είπατε ότι είναι πάρα πολύ δραστήριο, Θα είναι επαρκή όμω όλα αυτά που κάνει για να μπορέσουμε να επισπεύσουμε την πορεία μας. Και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω το εξή: Είπατε ότι ε, ότι εκατέρωθεν του Ατλαντικού έχουμε μία σκεπτικιστική κυβέρνηση. Ε, πώς μπορούμε να ε, το αντιμετωπίσουμε αυτό ε, οι στόχοι αηφόρου ανάπτυξη είναι κληροδότημα όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο και για τις μελλοντικέ μας γενναίες. Κύριε Στάινερ, αναφέρομαι ε, σε αυτό το ε, ψήφισμα της 6ης Ιουλίου του 2017 και λέγω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δείξει ότι, έναν πάρα, ότι είχε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ε, όσον αφορά την επίτευξη της αηφόρου ανάπτυξης όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ελπίζω να μην ήταν πάρα πολύ κακά τα αγγλικά μου. Ευχαριστώ. Okay, well, thank you very much. I was very tolerant. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είμαι μόνο επίκης μαζί σας επειδή είσαστε προσκεκλημένος στην Επιτροπή μας αλλά είμαι γενικώ επίκης ε, ε, με τους συναδέλφους. Μούσα Μούλη Μιάση από την Γκάμπια για να μας πει ορισμένα πράγματα για την ε, αντιπροσωπεία του και να ε, σχολιάσει όλα αυτά που είπε ο κύριος Σάινερ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι εδώ για να μοιραστώ μαζί σας αυτά που κάνει η χώρα μου η Γκάμπια προκειμένου να καλύψει τους ε, στόχους αηφόρου ε, ε, ανάπτυξης είναι θυμάμαι ότι το Δεκέμβριο του 2016 και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις του 2016 και 2017 ε, και τα αποτελέσματα των εκλογών είδατε ότι μπήκαμε σε μια νέα ε, περίοδο στην Κάμπια μας δίνει τη δυνατότητα να, να διατυπώσουμε τις αρχές μας και τους στόχους μας να αναβιώσουμε εθνικές πολιτικές ε, προσπαθώντας να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις και να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες του πληθυσμού πληθυσμού της Γάμπιας. Ο πρόεδρος της κυβέρνησής μας ε, προχώρησε στην ανάπτυξη της δημοκρασίας ε, σύμφωνα με το θεματολόγιο των στόχων του 2030. Η κυβέρνηση έκανε μεγάλα άλματα τα οποία μπορεί να καθοδηγήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τις πολιτικές που θα επιτρέψουν την παγκόσμια ειρήνη και την αηφόρη ανάπτυξη. Σε σχέση με το 2030 και τους σχετικούς στόχους για την αηφορία, η Γκάμπια ήδη πήγαινε ε. προς την επίτευξη των στόχων αυτών ε, ήδη από το 2000 και τη διακήρυξη των στόχων της χιλιετίας. Υπάρχουν βέβαια προκλήσεις. Ε, το κυβέρνηση, η κυβέρνηση δεν έκασε χρόνο. Κατήρτισε ένα νέο εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο εντόπισε τους τομείς προτεραιότητας της κυβέρνησης και να και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού. Ευθυγραμμίζεται με τους ε, στόχους ε, αηφόρου ανάπτυξης και έχει εθνικό και παγκόσμιο αντίκτυπο. Το σχέδιο τονίζει την ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση της ανάπτυξης, ε, εστιαζόμενο περισσότερο στις κλιματικές, στα κλιματικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα και τα ζητήματα ανισότητας. Επίσης, δεσμεύεται να καλύψει στόχους περιβαλλοντικής ε, αναβίωση του γεωργικού τομέα και βελτίωση της βιομηχανίας ε, προκειμένου να αναπτυχθεί η οικονομία. Η προτεραιότητα, οι προτεραιότητες της Γκάμπιας στο πλαίσιο αυτού του εθνικού σχεδίου ο κύριος στόχος καταρχάς θα μέσω των στρατηγικών προτεραιοτήτων. Ε, πρώτον, η αποκατάσταση της καλής διαχείρισης, ε, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, αποκέντρωση και τοπική αυτοδιοίκηση. Δεύτερον, σταθεροποίηση της οικονομίας μας, ε, μεταρρύθμιση της οικονομίας, αναδιαμόρφωση οικονομίας, εξυγχρονισμός της γεωργίας και της αλίας μας ε, για <coughs> καλύτερη διατροφή και επισητιστική ασφάλεια και μείωση της φτώχειας. Τέταρτον, επένδυση στους, στον πληθυσμό μας με τη βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών και τη δημιουργία μιας κοινωνίας πρόνοιας. Πέμπτον, ενεργειακές πηγές τις οποίες πρέπει να αποκαταστήσουμε για να υποστηρίξουμε την οικονομία μας και εκτών ε, ε, την πολιτιστική μας, ε, τη διατήρηση των πολιτιστικών μας μνημείων και να είναι κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης ο ιδιωτικός τομέας. We have seven Επτά εγκάρσιες ε, πολιτικές έχουμε που θα συμπληρώσουν τις στρατηγικές προτεραιότητες. Ε, πρώτον, ένας δημόσιος τομέας που θα είναι αποτελεσματικός και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Δεύτερον, η ενίσχυση των γυναικών της Γκάμπιας Λοιπόν, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό τους. Τρίτον, ενίσχυση της ε, διασποράς, ε, στην εθνική, της, διασποράς της Γκάμπια στην εθνική ανάπτυξη ε, καλύτερη χρήση της ε, γης και των αγροτεμαχίων, ε, να υπάρξει επίσης ψηφιοποίηση και να δημιουργηθεί μια σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, μια κοινωνία των πολιτών η οποία θα συμμετέχει στην εθνική ανάπτυξη και θα είναι συνεργάτης αυτής και απόφαση βάση επιστημονικών στοιχείων και στρατηγικών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ε, βέβαια και αλλαγή ε, του συντάγματος και ενίσχυση της αυτονομίας ε, των αυτο, πληθυσμών, ε, ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και ενίσχυση και επίσπευση της διαδικασίας απόδοσης δικαιοσύνης. Έχουμε επίσης αναμορφώσει τις γραμματείες μας ε, για να μπορέσουμε να ε, είμαστε πιο αποτελεσματικοί και υπάρχει ένας, δια, ένας μηχανισμός ε, μετάβασης και επαναπατρισμού και θα υπάρξει και μία νέα επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διερεύνησης της διαφθοράς. Θα ενισχύσουμε επίσης ε, την ε, υπηρεσία νομικής αρρωγής, ε, την υπηρεσία καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ανθρώπων, την ανεξαρτησία των εκλογικών επιτροπών και του Συμβουλίου Εθνικής Εκπαίδευσης. Έτσι θα μπορέσουν να είναι σε καλύτερη θέση να διεκπαιρεώσουν τα καθήκοντά τους βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και της μεταρρύθμισης της νέας κυβέρνησης. Όμως η βελτίωση των τομέων αυτών σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία και εταιρική σχέση σε διεθνές και εθνικό επίπεδο ε, το κατά πόσο η, θα μειωθεί, το, η μείωση της φτώχειας θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης ε, είναι σημαντικό κατά πόσο δηλαδή θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας και την επίτευξη των στόχων αηφόρου ανάπτυξης. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε συνάψει ε, με πολλές χώρες νέες ε, συμφωνίες, όπως με την Κίνα για παράδειγμα. Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενίσχυσης της, στον τομέα της ασφάλειας είναι πολύ σημαντική. Κάτι ακόμη που είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξή μας η ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης, η συμμετοχή στην κοινοπολιτεία, μια αμερόληπτη εθνική συνέλευση, μια η δημιουργία μιας επιτροπής συμφιλίωσης, η εξυγχρονισμός της ε, βιομηχανίας, η ανεξαρτησία του τύπου και ε, στρατηγικές ε, για την ασφάλεια και διακόπτη πρόεδρος. Συγγνώμη, μήπως μπορείτε να ολοκληρώσετε γιατί 4 κύριος Στάινερ. Αυτά είναι λοιπόν βασικά στοιχεία, συνεχίζει ο μιλητή, για τα οποία η Γκάμπια χρειάζεται υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους δωρητές. Τεχνική υποστήριξη δηλαδή και καθοδήγηση ενίσχυση την κυβέρ... της κυβέρνησης στη δημιουργία ε, ισχυρότερων θεσμών. Ευχαριστώ πολύ. Okay, Συνάδελφοι, θα είμαι πολύ πολύ αυστηρή με το χρόνο. Τρία άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Σας παρακαλώ πολύ ο καθένας όχι πάνω από 1,5 λεπτό. Και αν μπορείς να είστε και πιο σύντομοι, τόσο το καλύτερο γιατί έχουμε το αεροπλάνο. Ευχαριστώ πολύ Λίντα, ευχαριστώ πολύ κύριε Στάινερ για τις παρουσιάσεις όλων σας και τις προτάσεις σας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στρατηγικό πλάνο σε όλα τα επίπεδα εξάλλου, τοπικό επίπεδο και θα ήθελα να μας πείτε κάτι παραπάνω για αυτά τα εργαστήρια καινοτομία που δημιουργήσατε. Είναι μεγάλος ο κατακαιρματισμός από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει όμως μια πλατφόρμα που συντονίζει τα πάντα. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα, υπάρχουν διαφορετικές περιφέρειες και περιοχές πώς όλοι αυτοί επικοινωνούν και ανταλλάσσουν εμπειρίες και πληροφορίες. Είναι περίπλοκο το θέμα και όλοι αυτοί οι στόχοι σαφώς και είναι διαφορετικοί. Πείτε μου πώς κατανέμονται τα κονδύλια. Κάθε φορά χρειάζεται έλεγχος και είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς στην πολιτική, παραδείγματο χάρη στον τομέα της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης, κατανέμονται τα κονδύλια και πώς ελέγχεται η αποτελεσματικότητά τους. Και κάτι άλλο. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής το θέμα του περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουν όλοι αυτοί οι τομείς με αποτελεσματικότητα αν δεν υπάρχει ισότητα και δικαιοσύνη και ίση και δίκαιη ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ, Σεσίλ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω κύριε Στάινερ για τα όσα με είπατε, τα όσα συγκεκριμένα μας είπατε για να μας ενημερώσετε νομίζω ότι βεβαίως όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να κατευθυνθούμε προς μια βιώσιμη αερφόρο ανάπτυξη με επί τη βάση του προγράμματος τούτου και πώς θα πούμε όλα αυτά τόσο γρήγορα αλλά θα πρέπει να καλύψουμε όλα αυτά τα ζητήματα που είναι αλληλένδετα και τα οποία δεν πρέπει να κανείς να τα βλέπει ξεχωριστά. Χρειάζεται επομένω συνολική σφαιρική προσέγγιση, τέτοια παγκόσμια ε, προσέγγιση και σε κοινωνικό επίπεδο, να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούν τους ανθρώπινους ε, πόρους και για πέστε μας πώς θα γίνουν αυτές οι επενδύσεις από τις κυβερνήσεις με τα διάφορα μοντέλα, όλοι οι θεσμοί αυτοί που θα πρέπει να επιστρατευθούν ούτω ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτούς τους ε, στόχους, άρα ανθρώπινοι πόροι. Εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε. Ε, στον άνθρωπο. Αυτό το πρέπει να είναι το επίκεντρο. Παραγωγικά μοντέλα τα οποία να είναι συμβατά με τους 17 στόχους, με όλους τους 17 στόχους της ε, αηφόρου και επίσης να επισημάνουμε τα μοντέλα για την καλύτερη εκβιομηχάνηση, τον εξυγχρονισμό και θα πρέπει επίσης να δούμε αυτό το οποίο είπαν τόσοι. Να πρέπει αυτό να μην το παραβλάψουμε. Το περιβάλλον. Έχουμε την μπλε οικονομία, την πράσινη οικονομία, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά όλα αυτά χωρίς σφαιρική συνολική προσέγγιση δεν βγαίνει. Και επίση να λάβουμε υπόψη και αυτά που είπαν από την ε, Γκάμπια. Θέλουμε δημοκρατία της ειρήνης και αυτό να το πετύχουμε με τις διάφορες συμφωνίες. Ναι, προσέγγιση από τη βάση αλλά να τηρηθούν τα όσα προβλέπει το θεματολόγιο του 2030. Έλλη. Ε, ευχαριστούμε που ήρθατε και που μας τονίσατε πόσο σημαντική είναι αυτή η στόχη. Αν θα πρέπει όλα να τα λάβουμε υπόψη και να τα συγκεράσουμε. Να λάβουμε υπόψη τους πάντες και τα εθνικά κοινοβούλια, τις τοπικές αρχές, Κανείς δεν μείνει απ' έξω. Αυτό θα μας εγγυηθεί το ελεύθερο μέλλον και αυτό από τα πρώτα βήματα με το που εγκρίθηκε αυτό το θεματολόγιο ξεκίνησε η προσπάθεια. Πότε θα πρέπει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και κομισιό να βρουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ε, επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των σχετικών στόχων. Είπαμε ότι οι διαδρομοί ξεκίνησαν από το 2015, αλλά πολλά άλλαξαν έκτοτε. Και πολλά άλλαξαν προς το χειρότερο. Και μερικές χώρες πήραν το στραβό δρόμο λόγω αλλαγής κυβέρνησης, όπως η Θα πρέπει να δούμε επομένω ποιοι είναι παράδειγμα προ μίμηση για αυτού του στόχου που είναι τόσο φιλόδοξοι. Δεν πρέπει αυτά να μείνουν νεκρό γράμμα. Και θα μείνουν εάν δεν διαθέσουμε αρκετή πληκότητα. Επομένω η Ευρώπη θα πρέπει να προσπαθήσει το 0,7% να το πετύχει. Πώς το λένε, πώς το λένε. Α, το, το ΑΕΠ, το ΑΕΠ, ναι, ναι, ναι. Α, και να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την φουσκωμένη ενίσχυση. 0,26 είναι στην Ιταλία. Αλλά αν βγάλουμε τις δαπάνες για τους πρόσφυγες στην Ιταλία, ε, η φύρα είναι το 0,20. Άρα θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τοπικούς εθνικούς πόρους για να μπορέσουμε να καταπολέμησουμε την φορά αποφυγή και επίση και το πώς να μην φεύγουν οι μας να πηγαίνουν ξέρω εγώ στην Αφρική. Α, ναι, ευχαριστώ που μου το είπατε. Δεν αρκεί αυτό το, το, το, το το ΑΕΠ ως κριτήριο δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με αυτό το κριτήριο η ανισότητα. We're discussing, um... Τώρα έχουμε λίγα λεπτά για τις απαντήσεις. Ξέρετε βεβαίως ότι η στόχοι αυτή είναι πολύ και δεν ανταποκρίνεται όλοι σε αυτά που ρωτήσατε. Ο κύριος Στάινερ. Όπως είπα από την αρχή, δεν πρόκειται για τη μόνη στιγμή που θα συζητήσουμε για τα θέματα αυτά. Δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος αυτής της συζήτησης που έχουμε. Οι συνάδελφοι από την Αφρική έφυγαν, αλλά πραγματικά η συζήτηση, αν θέλετε, μεταξύ Ηνωμένων Εθνών και Κοινοβουλίου συνεχίζεται. Το θέμα της λογοδοσίας φυσικά ξεκινάει ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Το θέμα είναι ότι η εκτελεστική εξουσία, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών έχουν συγκεκριμένους ε, κανόνες που αφορούν τη διαδικασία της λογοδοσίας, της αξιολόγησης, της προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων κτλ και τα εθνικά κοινοβούλια βεβαίως έχουν το ρόλο τους, αλλά σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις νομοθεσίες και από την ρύθμιση που προβλέπεται στη κάθε χώρα. Βεβαίως ε, η Διεθνής Ένωση Κοινοβουλίων είναι κάτι είναι πολύ ενδιαφέρον και σε όλα τα επίπεδα η κοινοβουλευτική συνεργασία σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σίγουρα μπορεί να προσθέσει ε, μία διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, οι πολίτες της Ευρώπης είναι πολύ δραστηριοποιημένοι όσον αφορά τους ε, στόχους αυτούς τους αναπτυξιακούς αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξέρω, οργανώνεται ακροάσεις. Σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσετε να βάζετε στο επίκεντρο της εργασίας σας τους στόχους και αυτό είναι η μία διάσταση. Είναι πολύ χρήσιμο όταν το κάνετε αυτό. Μίλησα για τις πλατφόρμες, μίλησα για τη διμερή συνεργασία αλλά και για την στρατηγική αυτή που βάζει στο, στην καρδιά των επενδύσεων τους αναπτυξιακούς στόχους. Σημασία έχει να υπάρχει συνοχή, να υπάρχει συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά τα επενδυτικά προγράμματα. Το οικονομικό παράδειγμα είναι σημαντικό το μήνυμα που περνάμε, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε μεγάλο βαθμό νιώθουν παραμερισμένοι, εγκαταλελειμμένοι και απομονωμένοι. Και αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις για τη δημιουργία υποδομών, για τις επενδύσεις, για την ανάπτυξη, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό. Οι επενδύσεις είναι αποτελεσματικές όταν δεν χάνουμε ε, από το κέντρο μας όλες αυτές ε, τις προτεραιότητες. Πέρσι είχαμε 48 χώρες που πραγματικά συμμετείχαν και 60 που θέλουν φέτος να κάνουν ε, ε, έκθεση, να υποβάλουν προτάσεις. Αυτή λοιπόν η στόχη είναι ένας πολλαπλασιαστής, ένας παράγοντας επιτάχυνσης και ανάπτυξης και συσπήρωσης προτάσεων και επενδυτικών ε, ε, προγραμμάτων σε τεράστιο βαθμό. Πολλοί έχουν εκφράσει βέβαια και ανησυχίες και επιφυλακτικότητα. Αλλά αυτή η επιφυλακτικότητα πολλές φορές δημιουργεί και μία ε, δυσκολία, αποσταθεροποίηση. Κοιτάξτε παραδείγματο χάρη τι γίνεται σήμερα με τους Παλαιστινίους. Κοιτάξτε τι γίνεται με τους πρόσφυγες. Η αποσταθεροποιητική, αν θέλετε, διάσταση αυτού του φαινομένου είναι τεράστια. Και όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Σημαντικό είναι να δούμε πώς θέλουμε να προωθήσουμε αυτές τις αναπτυξιακές επενδύσεις. Πώς επενδύουμε εμείς οι ίδιοι στις δικές μας κοινωνίες και πώς επενδύουμε οι μεν στις προτάσεις, στα προγράμματα και στις υποδομές άλλων χωρών. αυτού του είδους οι επενδύσεις δεν πρέπει να διακατέχονται από ανταγωνισμό, από ανταγωνιστικότητα, αλλά από αλληλεγγύη. Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να μας καθοδηγήσει. Και με αυτόν τον τρόπο περνάμε σε κάποιους τομείς που φαίνονται αδύνατο να τους διαχειριστούμε, που φαίνεται αδύνατο να τους χρηματοδοτήσουμε και που φαίνεται αδύνατο να τους οραματιστούμε. Χρειάζεται αμοιβαία συνεργασία. Ο Γενικός Γραμματέας μιλάει για την δήλωση της ε, συνεργασίας που είναι απαραίτητη, της αλληλεγγύης και της αλληλοεξάρτησης. Βλέπω πολλά φιλικά και γνωστά πρόσωπα σε αυτή την αίθουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Πραγματικά αυτό το κοινοβούλιο έχει δείξει πολλές φορές την αλληλεγγύη του και το πόσο πιστεύει στα πολυμερή προγράμματα. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλό ταξίδι. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρχουν ε, απεργίες που θα σε εμποδίσουν να φτάσετε γρήγορα στο αεροδρόμιο.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 εδώ απηχούμε τις απόψεις του. Και αυτό θα κάνω κι εγώ. Αλλά δεν θα με γρηγορήσω. Λίγα λεφτάκια μόνο θα σας τα πω. Είναι γνωστό ότι <clears throat> από με τι εξωτερικής πολιτικής που έχει η ευρωπαϊκή πολιτική ε, η Επιτροπή ε, ε, Ανάπτυξης συνδέεται με τρία από αυτά τα μέσα όσον αφορά πρώτα το εργαλείο αναπτυξιακή συνεργασία, το Ταμείο Ανάπτυξης αλλά επίσης και το Ταμείο Ανθρωπιστικής Δράσης. Και εμείς ασκούμε έναν κυλευτικό έλεγχο, λέγω έλεγχο, με διάφορες ομάδες εργασίας όσον αφορά αυτό το μέσο αναπτυξιακής εργασίας και ταυτόχρονα έχουμε διαρθρωμένους διαλόγους με την Επιτροπή για κάποια στρατηγικά θέματα και για το περιεχόμενο των πολιτικών της Ένωσης. Οπότε ο στόχος της έκθεσης είναι το να βάλω το λιθαράκι μου εις την τροποποίηση αυτών των τριών μέσων πολιτικής που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δούμε πόσο δόκιμα αυτά τα μέσα σε σχέση με τους στόχους που ετέθησαν όταν αυτά τα μέσα επενοήθησαν. Και να εξετάσουμε πώς ε, λειτουργήσαν από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο του 2017. Επίσης, η έκθεση προσπαθεί να καταδείξει το τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτές τις εκθέσεις μέχρι το της διαδρομής τους, δηλαδή το 2020 και τι είδους προτάσεις, ε, ιδέες, συστάσεις μπορούμε να σκαρφιστούμε για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αρχάς του 21 δηλαδή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να παρουσιάσει το Μάιο κάποια στιγμή την πρώτη της πρόταση για αυτό το επόμενο πι δέλτα πι. Η έκθεση έχει λάβει υπόψη τη σχετική τεκμηρίωση βάση εξολογήσεων άλλων θεσμικών οργάνων και βασικά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, κάποιες ΜΚΟ, κάποια συνδικάτα και επίσης και επί τη βάση των όσων πρότεινε το κέντρο τεκμηρίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο που μας βοήθησε ούτως ώστε να κάτσουμε και να δούμε αυτές τις εξωτερικές αξιολογήσεις. Η έκθεση. Βασικά σημεία έχει τα εξής. Πρώτα πρώτα. Λέμε ότι με θα υπέρ του να παραμείνει ή να αυξηθεί η ενίσχυση της αντισιακής βοήθειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι πιο εκτεταμένο και θα είναι και πιο σημαντικό για το μέλλον, γιατί διάφοροι διεθνείς παίκτες, όπως είπα τώρα, έχουν προβεί σε περικοπές ή έχουν κλείσει τελείω τη στρόφιγγα για το πόσα εισφέρουν σε διάφορους τομείς της αμυσιακής βοήθειας. Ε, επίσης, λέμε ότι είμεθα υπέρ του να διατηρηθεί η ταυτότητα, η μοναδικότητα αυτών των στόχων, των αξιών, των αρχών της αμυσιακής βοήθειας και της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας και να δούμε πώς δεν θα υπάρξει χειραγώγηση, εκμετάλλευση, καπέλωμα αυτών των πολιτικών στην εξωτερική πολιτική. Ούτε να έχουμε τίποτε λαθροχειρίες και να πάνε οι πόροι της ανάπτυξης αλλού, σε άλλες πολιτικές ένωσες. Που θεμητή είναι η αλλά δεν μπορεί να παίρνουν πρικοδότηση της ανάπτυξης. Επίσης λέμε ότι και για τώρα και για το μέλλον θεωρούμε ότι η διεθνή συγκυρία άλλαξε από το 2014 που εγκρίθηκαν αυτά τα μέσα πολιτικής. Άλλαξε το θεματολόγιο της βιώσιμης ανάπτυξης, άλλαξε το θεματολόγιο της ε, Αντισαμπέμπα, το πλαίσιο Σεντάι για τις καταστροφές, η ανθρωπιστική κορυφή της Κωνσταντινούπολης, η κλιματική κορυφή του Παρισιού. Ε, λοιπόν, να, και για τη δική μας δράση έχουμε την έγκριση της παγκόσμιας πολιτικής για την ε, ασφάλεια. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την ανθρωπιστική βοήθεια και την άλλη γενικότερη σύνδεση που έχει διαμορφωθεί για πολιτική και ανάπτυξη. Και άρα σε αυτό το καινούργιο τοπίο θα πρέπει να κινηθούμε και να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Και τώρα για να αξιολογήσουμε τα διάφορα από αυτά τα εργαλεία και μέσα λέμε ότι καταρχήν ε, και η αναπτυξιακή βοήθεια και το Ταμείο για την Ανθρωπιστική βοήθεια έχουν προσαρμοστεί γενικώ σε αυτά που έπρεπε να κάνουν όταν επινοήθηκαν έχουν κινηθεί στα πλαίσια ε, των κανόνων λειτουργίας τους με κατεύθυνση την βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης καταφέραμε σε έναν σημαντικό βαθμό να συγκρατήσουμε τη φτώχεια στον κόσμο που είναι βασική αρχή της πολιτικής μας για την αντιστοιχική βοήθεια. Αναχαιρετήσαμε, βοηθήσαμε σε διαφορετικές κρίσεις στον κόσμο και κινηθήκαμε με ευελιξία, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε αποδεκτή, αρκετά καλή επιτυχία. Τώρα για την εμπιστιακή βοήθεια, του συγκεκριμένο εργαλείο πολιτικής, που καλά λειτουργήσε όσον αφορά την ευελιξία, καλά λειτουργήσε όσον αφορά το θεματικό πρόγραμμα και η εκτέλεση διέπεται από κάποιους μηχανισμούς ε, κάπως γραφειοκρατικούς, δηλαδή αργούμε, αργούμε να επέμβουμε επί τόπου. Οπότε στην έκθεση λέμε ότι ανησυχούμε γιατί έπρεπε να τουλάχιστον 20% των ενισχύσεων της ε, αναπτυξιακής βοήθειας να έχουν διατεθεί για παιδεία, δευτεροβάθμια και τις βασικές υπηρεσίες ενίσχυσης περισσότερη πρικοδότηση και επίσης λέμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και στο τέλος ίσως από το 16 και μετά αυτό το Ταμείο Ανάπτυξης όπως ξέρουμε το διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη και αιτήσει των κρατών μελών Έπρεπε το Ταμείο να αντιμετωπίσει όλα και περισσότερες ανάγκες για ασφάλεια, μετανάστευση. Οπότε πολλές φορές θα έπρεπε να συμβιβαστούμε όσον αφορά την τήρηση βασικών αξιών. Τώρα όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια μπορέσαμε με ευελιξία και επειδή συχνά υπήρχε προοικοδότηση εξαιρετική να καλύψουμε πολλές κρίσεις σε όλο τον κόσμο και το πρωί είδαμε το πώς καταφέραμε να υπάρχει μια σόρευση καλύψεων, σόρευση παρεμβάσεων, παρά το ότι οι ανάγκες ήταν πάρα πολύ πιστικές Μπορέσαμε δηλαδή να βοηθήσουμε όλους εκείνους όπου και αν βρισκόντουσαν εκείνους που χρειαζόντουσαν την αραγή μας. Τώρα όσον αφορά τις συστάσεις για την ε, υπόλοιπη περίοδο, δηλαδή μέχρι το 2020, στην έκθεση λέμε ότι θα πρέπει να μην υπάρχει κατάχρηση των καταπιστευμάτων. Μια που τα κράτη-μέλη, τα οποία όταν ε, φτιάξανε αυτά τα καταπιστεύματα, δεσμεύονται, αλλά δεν εισφέρουν όσα δεσμεύτηκαν. Οπότε όλα αυτά παραβλάπτουν την προσπάθεια και την πολιτική της αναπτυσιακής συνεργασίας. Τέλος πάντων. Όπως πάντα επιμένουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια σε αυτά τα καταπιστήματα, οπότε και το Κοινοβούλιο στα πλαίσια του οικονομικού ελέγχου εποπτεύει αυτά τα καταπιστεύματα βέβαια έχουμε τόσες κρίσεις που θα πρέπει να καλύψουμε μέχρι το 2020 οπότε και αυτά όλα τα μέσα να επιδείξουν ευελιξία. Να διέπονται από ευελιξία ούτως ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι αποθεματικά υπάρχουν που προλάβονται για αυτές τις κατεπιστές περιπτώσεις και επίσης ζητούμε ότι το, ο μηχανισμός ανθρωπιστικής βοήθειας να χρησιμοποιηθεί ακριβώς σύμφωνα με όσα έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην συνάντηση της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, φυσικά και λέμε θέλουμε να γνωριστεί η ιδιωτυπία της ανθρωπιστικής βοήθειας και αν ζητηθεί συγκεκριμένη ε, αντιμετώπιση της ε, βοήθειας θα πρέπει και αυτή να ανταποκρίνεται στην ένταση των αναγκών. Τώρα, για την περίοδο μετά το 2020 θέλουν να είναι αυτόνομε αυτέ οι πολιτικές ανάπτυξη και τη ανθρωπιστική βοήθεια, θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε την, την, ιδέα, το ότι μέσω της ε, συνεργασία μα και τη ανθρωπιστική βοήθειας η Ένωση να προβάλλει περισσότερο την εικόνα τη ω παγκόσμιο παίκτη. Soft power όπω το λέμε. Δηλαδή ένα ε, παράγον που να είναι αποτελεσματικό για τι συγκρούσει για την επίλυσή τους, για την ειρήνευση μέσα από τέτοιες πολιτικές. Και φυσικά να αυξηθεί και η επίσημη πρικοδότηση για την ανάπτυξη. Γιατί τώρα ιστερεί σε σχέση με τα όσα έχουμε υποσχεθεί, με όσα δηλώσαμε ότι δεσμευόμαστε να παράσχουμε. Επίσης, αναδεικνύουμε το ότι ή στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε βελτίωση των επιδοσιών μας στην απλούτευση και ευελιξία. Όμως τούτο δεν μπορεί ποτέ να είναι εις βάρος του ελέγχου, του συνομοθέτη δηλαδή του κοινοβουλίου μας. Τώρα αφορά την ε, ένταξη του Ταμείου Ανάπτυξης, εμείς ανέκαθεν είμεθα υπέρ αυτής της ένταξης της ε, ένταξης στον προπολογισμό δηλαδή. Έτσι θα πετύχουμε περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη συνέπεια στην πολιτική της ανάπτυξης. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει με την ένταξη στον προπολογισμό να χαθεί η νομιμοποίηση και ο δημοκρατικός έλεγχος από Βουλάς κοινοβουλίου. Εν Σας τονίζω τα εξής η έκθεση. Αρχικά αφορά την υλοποίηση της πολιτικής ανθρωπιστικής ενίσχυσης και ανθρωπιστικής βοήθειας. Όλα αυτά σε μια συγκυρία, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει τις προτάσεις για το 2020. Άρα πρόκειται για μια ευκαιρία. Μπορεί η Επιτροπή μας να εκφράσει τις απόψεις της πώς θέλουμε να εφαρμοστούν αυτά τα μέσα πολιτικής ε, μέχρι το τέλος της διάρκειας ζωής τους. Και άρα θέλουμε επιτροπή. Όταν παρουσιάσει τις προτάσεις δηλαδή τον Μάιο, για το επόμενο πι θέλτα πι, να μας πει τι μέσα θα μετέλθει. Να αναδειχθεί η μοναδικότητα η ιδιοτυπία τέλο πάντων ανθρωπιστική βοήθεια και συνεργασία για την ανάπτυξη. Τελευταία παρατήρησή μου είναι η, η επιτροπή μα πρέπει να τοποθετηθεί αφού η Κομισιόν το Μάιο παρουσιάσει τι προτάσει τη. Και έτσι να τοποθετηθούμε αλλά να τοποθετηθεί και η καινούργια Επιτροπή Ανάπτυξη μετά τι ευρωεκλογέ του 19. Μα δεν είναι δυνατόν ένα κοινοβούλιο που θα εκλεγεί τον Μάη του 19 να μην πει τίποτα όσον αφορά το πι δελτα που θα καλύψει αυτά τα ε, μέτρα, αυτά τα μέσα πολιτικής τέλο πάντων, τα οποία θα αρχίσουν να τρέχουν πρώτη πρώτη του 21, δηλαδή σχεδόν 1,5 χρόνο μετά την αρχή της θητείας του. Άρα θα πρέπει να προβλέψουμε τι θα γίνουν τα προβλήματα στο μέλλον και, παράλληλα να χαράξουμε την πορεία. Μια πορεία που είναι πάρα πολύ βασική για το ρόλο του Κοινοβουλίου στην ανάπτυξη. Ναι. και ταυτόχρονα θέλω να πω στου και ηγητές ότι παρακαλώ μην θέλετε να ξαναεφεύρετε τον τροχό ε, ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο και με άλλους τρόπους, όχι μόνο με το δικό μου κείμενο και με άλλα που το κάνουμε. Ευχαριστώ Ενερίκη, που μας έκανες μια τόσο καλή απεικόνηση της κατάστασης και μας έδωσε τόσο καλές κατευθυντήριες γραμμές. Πάντα λέω στους συναδέλφους, αν δεν υπάρχει ένα, ένας πραγματικός λόγος και ένα πραγματικό μήνυμα, μην υποβάλλετε τροπολογίες, γιατί χάνετε το βασικό μήνυμα. Οπότε καλό είναι να συντονίζουμε τις απαντήσεις μας και αν θέλουμε να απευθύνουμε ένα βασικό μήνυμα σε άλλα όργανα να μην έχουμε ε, χιλιάδες επί χιλιάδων ε, τροπολογίες. Ε, πρώτα ο Φρανκ Έγκλ από το ΕΛΚΑ, πρώτος της εισηγητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω ούτε να ε, σκοτώσω το προϊόν, το προϊόν σου, φίλε Ενρίκε, δεν ε, θέλω να σε δυσαρεστήσω. Όμως, ε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι μία προσέγγιση που επί της οποίας, επί της οποίας είμαι σύμφωνος όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία ε, υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία για τα οποία θα καταθέσω τροπολογίες γιατί δεν συμφωνώ απολύτως με την προσέγγιση σου. Για κάποια στοιχεία, μία στάση που τη βρήκα κάπως επιφυλακτική όσον αφορά την ε, βοήθεια την ε, δημοσιονομική. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεπεράσουμε τον αναπτυξιακό πατερναλισμό και να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό ε, μέσω της αναθεώρησης της ε, δημοσιονομικής βοήθειας. Να μην το κάνουμε δηλαδή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το κάνουμε αυτό ας πούμε στην Κεντρική Αφρική γιατί αν και κανένα κριτήριο δεν ε, πληρούνται γιατί πρέπει να πληρώνει τους στρατιώτες της, τους υπαλλήλους τους. Αν δεν υπάρχει τίποτε στον προπολογισμό της χώρας, δεν θα, μπορούσαμε να, δεν θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να πληρώσουν τους υπαλλήλους τους και τους στρατιώτες τους. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσω μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης. Πρέπει λοιπόν να το αποδεχθούμε αυτό, να αποδεχθούμε λοιπόν ένα μέσο το οποίο δεν θα ήταν κατά τα άλλα σε άλλες περιπτώσεις όριμο όμως πρέπει να αποδεχθούμε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι εταίροι μας στον κόσμο γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι επιμένουμε ότι δεν ε, καταφέρνουν τελικά να διαχειριστούν μόνοι τους τη χώρα τους. Άλλο είναι ο ανταγωνισμός στην, ε, ε, στην ανάπτυξη. Αν θέλουμε δηλαδή να αντιταχθούμε στην Κίνα, στη Ρωσία, στην Ινδία, στη Βραζιλία και σε άλλες χώρες που διαφαίνονται ως ανταγωνιστές, ε, σε σχέση με τα συμφέροντά μας στον κόσμο της ανάπτυξης πρέπει η στάση της Ευρώπης ε, όχι μόνο να την πάρουμε σοβαρά αλλά να θεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο ότι αξιοποιεί την ε, την προσπάθεια των κρατών μέλων. Σίγουρα θα βρούμε διατυπώσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να λύσουμε αυτή την μικρή μας διαφορά. Συμφωνώ με όλα αυτά που είπες και τα εκτιμώ ιδιαίτερος όσον αφορά την ε, ε, ευελιξία, την απλοποίηση, τη δημιουργία αποθεμάτων ε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο όταν θα είναι απαραίτητο, γιατί νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ανταποκρινόμαστε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τώρα. Υπάρχει δηλαδή μια άμεση ανταπόκριση ταχύτερη σε σχέση με την τωρινή, ε, γιατί είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως χρειάζεται και πάλι στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Οι Κινέζοι φίλοι μας ε, είναι πιο γρήγοροι από μας. Αύριο οι Τούρκοι, άλλοι, μεθαύριο άλλοι. Γιατί, γιατί είμαστε πολύ διαδικαστικοί. Γιατί χανόμαστε μέσα σε χιλιάδες ομάδε τυπικότητες, ενώ οι άλλοι έχουν ήδη αναλάβει δράση. Αυτό πραγματικά νομίζω μας ε, ε, στοιχίζει σε γόητρο και ε, σε σεβασμό. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Επιβεβαιώνοντας ότι η δική μου ομάδα θα είναι βεβαίως διαθέσιμη για να τελεσφορήσει όλη αυτή η διαδικασία, γιατί έχει σημασία με ολόκληρη τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλο τον κόσμο. Η δράση μα υπέρ τη ανάπτυξη είναι ένα σημαντικός παράγον αυτής της αξιοπιστίας Ευρώπη. Ευρώπης. Ε, συνεπώς, όντω πρέπει να εμπλακούμε με πολύ αποτελεσματικό, ε, τάχιστο τρόπο, ειδικότερα στι περιπτώσει ανθρωπιστική βοήθεια, ανθρωπιστικών κρίσεων. Συγγνώμη. Αυτό είναι προ όφελο όλων μα, προ συμφέρον όλων μα και είναι προ συμφέρον όλων μα να λειτουργήσει και καλά. Οπότε φυσικά θα σε υποστηρίξουμε στο κείμενό σου. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Η Σεσίλ Κιέγγε. Ενρίκε, ευχαριστούμε για τόσα σημαντικά μας είπες με την έκθεσή του για την εφαρμογή αυτών των μηχανισμών. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά μας δίνουν να καταλάβουν πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι μηχανισμοί. Ε, συνεργασία αναπτυξιακή, ανθρωπιστική βοήθεια, βοήθεια για την ανάπτυξη. Εγώ τώρα θέλω να επικεντρώσω την προσοχή μας σε κάτι άλλο. Κάτι που σκέφτηκα σε μια αποστολή στην Αφρική. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, πολύ καλά τα λες Ενρικέ, αλλά απαιτούν κάποια κριτήρια. Κάποιε μεταβλητέ, κάποια χαρακτηριστικά, όπω η ευελιξία που μα είπες. Αλλά αυτό αφορά και τα κατεπίγοντα καταπιστεύματα. Θα πρέπει όλοι αυτοί οι μηχανισμοί να είναι βάση για την πολιτική ανάπτυξη. Ολοκλήρωσαν κάποια διαδρομή και έχουμε τις συμφωνίες DCI όπως τα συζητήσαμε πριν από λίγες μέρες και προσπαθούμε να δούμε τι μορφή θα πάρει αυτή η μεσοπρόθεσμη αξιολόγησή μας. Όλα αυτά τα λέμε για να δούμε τι είδους αξιολόγηση θα κάνουμε όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί με βοήθησαν ξεκάθαρα να διαπιστάσω το πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη λογική που διέπει αυτούς τους μηχανισμούς. Και με τον ε, συναδελφό Βέντα πήγαμε στη Σενεγάλη και είδαμε για ε, τα καταπιστεύματα πώς λειτουργεί η υπόθεση. Μια ολόκληρη μέρα με αυτό ασχοληθήκαμε και επομένως όλοι αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει να αποκτήσουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό, την αντοχή. Αυτό να αναβαθμίσουμε, να αλλάξει άρα η προσέγγιση μας, να μπορέσουμε να αναδείξουμε τους ανθρώπινους πόρους, τον άνθρωπο. Αυτό θα έχει αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη πολλών χωρών. Με αυτονομία μια που πολλές από τις εν λόγω περιοχές με τις οποίες εργαζόμαστε θα πρέπει να κατευθυνθούν προς την αξιοποίηση των νέων πόρων. Μέχρι τώρα η λογική μας είναι η λογική της ενίσχυσης, μονόδρομος. Χρειάζεται εταιρική σχέση win-win. Ε, πού να τη βρούνε στην αυτονομία. Άρα, αναθεώρησε υπό το φως των όσων συμφωνήσαμε στο Αμπιτζάν. Νέα προσέγγιση. Και θα ήθελα το Κοινοβούλιο, αλλά σίγουρα και η Κομισιόν, να αλλάξουν ρότα και να ενισχύσουν αυτή την ανθεκτικότητα. Και έτσι σε τοπικό επίπεδο ο κόσμος σιγά σιγά να μπορέσει να πετύχει την ανάπτυξη. Με αυτονομία. Και ταυτόχρονα να καταπολεμηθούν οι διάφορες ρίζες προβλημάτων που αποτελούν φραγμό στην ευημερία του κόσμου. Αυτό θα είναι ένας θετικός καταλήτης, αυτό θα είναι κίνητρο για την ε, ντόπια ανάπτυξη. Μαρία Χόιμποκ. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία Χόιμποκ. Ευχαριστώ πολύ. Η Χάιντι Χαουταλά δεν είναι σήμερα εδώ και την ε, αντικαθιστώ όσο μπορώ βέβαια. Χαιρετίζουμε τη γενική κατεύθυνση αυτής της έκθεσης. Πιστεύουμε όμως ότι πρέπει να τοποθετηθούμε με σαφήνεια. Διαφορετικά εργαλεία ανάπτυξης από αυτά της ανθρωπιστικής ε, ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι χρειάζονται αξιόλογοι τρόποι, συγγνώμη, τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε αξιολογήσεις, με τους οποίους μπορούμε να μετρήσουμε σωστά και να ελέγξουμε οι αξιολογήσεις, είναι σημαντική καθότι πρέπει να είναι στοχευμένα τα εργαλεία και τα μέσα. Ένας από τους ε, κριτές, ένας από, τους, από τις παραμέτρους που θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου είναι εάν η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους, εάν υλοποιούμε αυτά που είχαμε θέσει αρχικά σαν στόχους. Λυπούμαστε ιδιαίτερα γιατί δεν έχει αξιολογηθεί το Africa Peace Facility, ενώ χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια. Επίσης βλέπουμε ότι έχουν προκύψει δυσκολίες και προβλήματα, κάτι που έχει πλήξει την αξιοπιστία της δράσης και την το κατά πόσο η χρήση των κονδυλίων γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο. Πρέπει λοιπόν εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πολύ πιο αυστηρή και προσεκτική. Yeah, thank you. And uh, just maybe... Ευχαριστώ. Να προσέξω και εγώ το όνομά μου στον κατάλογο των ομιλητών. Είναι πολύ καλή η έκθεση αυτή. Συμφωνώ με όλα που παρουσίασες. Αυτά που είπε ο Φρανκ Έγγελ όσον αφορά τους τομείς που πολλές φορές ξεχνάμε. Μιλάμε για ανταγωνιστικότητα και μιλάμε και για ανταγωνισμό στην Αφρική χωρών που προτείνουν τη βοήθεια και την αναπτυξιακή συγκεκριμένα βοήθεια. Εμείς είμαστε αργοί. Έχουμε βαριές διαδικασίες. Κάτι πρέπει εδώ να σχολιάσει η Επιτροπή. Θυμάμαι πριν από χρόνια ήταν ε, ο Νίλ Κίνοκ επίτροπος και μιλούσαμε τότε για τα σχέδια, για τον τρόπο αξιολόγησης και ανησυχούσαμε για το πώς θα αξιολογηθεί η δράση μας εκεί. Λέγαμε μάλιστα ότι πρέπει να μην ε, είμαστε ρηψοκίνδυνοι. Πιστεύω ότι πρέπει όμως αντίθετα να τολμήσουμε, να δείξουμε φαντασία, δημιουργικότητα. Λίγα χρήματα χρειάζονται και πολλές ιδέες. Ιδέες που θα οδηγήσουν σε επιχειρηματικότητα ή όχι απαραίτητα σε επιχειρηματικότητα. Πολλές φορές χρειάζονται πολύ μικρά ποσά, μικροπιστώσεις. Θυμάστε χτες η ομιλήτρια από τη Γερμανία η οποία μας έδωσε τα παραδείγματα όλων αυτών που παίρνουν ένα μικρό δάνειο και αποτυγχάνουν. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και στις χώρες μας. Ναι, γιατί να μην αποτυγχάνουν και εκεί. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει ένα σωστό επιχειρηματικό μοντέλο και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουν. Μιλάμε όμως πολλές φορές για σχέδια που χρειάζονται μικρά ποσά, λογικά ποσά. Οι κίνδυνοι λοιπόν που πρέπει να αναλάβουμε και να στηρίξουμε θα πρέπει να είναι υπολογισμένοι, ελεγχόμενοι και λογική. Αλλά παραδείγματος χάρη αυτόν που συναντήσαμε με αυτό το μηχάνημα που ξεφλωδίζει τα φιστίκια ήταν μια πολύ έξυπνη ιδέα ήταν ένας έξυπνος νέος ο οποίος είχε αυτή την ιδέα και μόνος του κατασκεύασε μία μηχανή. Αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον στηρίξουμε και τα χρήματα που χρειάζονται είναι ελάχιστα. Αλλά βέβαια χρειάζεται ένα συντονισμός και τελικά υπάρχουν και όλα τα επίπεδα των ελέγχων, των διαδικασιών που εκεί χάνονται πολλά χρήματα. Όντως λοιπόν Πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μας, γιατί συνεχίζουμε να είμαστε ο πιο σημαντικός χρηματοδότης. Είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής και αυτό μην το ξεχνάτε. Και πολλές φορές οι εταίροι μας, αυτοί που συγχρηματοδοτούν τα προγράμματα μαζί μας, ίσως είναι πιο κοντά στη δράση, πιο κοντά και ίσως η προστιθέμενη αξία τους είναι άλλη. Είναι ότι μπορεί πολλές φορές να γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση. Χρειάζεται λοιπόν και εμείς να ξαναδούμε λίγο τον τρόπο λειτουργία μας. Η Επιτροπή είναι εδώ. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή καταρχήν. Πρόκειται για ένα σχέδιο που πραγματικά καλύπτει πολύ ενδιαφέροντα και πολλά σημεία τα οποία τα παρουσιάζει εξάλλου με πάρα πολύ ισορροπημένο τρόπο. Βεβαίως στα πλαίσια του πολιετούς χρηματοδοτικού πλαισίου και στην προετοιμασία του νέου πλαισίου το θέμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Θα κάνω τρία σχόλια το πρώτο ενδεχομένως απαντάει και μία από τις ερωτήσεις στην παράγραφο 10. Το θέμα δηλαδή του σεβασμού, του στόχου του 20% των κονδυλίων που θα πρέπει να αφιερώνονται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, συνεργασία δηλαδή στην ανάπτυξη αυτό το 20% το τηρούμε, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Ο στρατηγικός διάλογος που θα γίνει στις 6 Μαρτίου για τη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση, νομίζω ότι αν σας ενδιαφέρει θα μπορούσαμε με αυτή την ευκαιρία να σας δώσουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία αριθμητικά για να δείτε ότι τηρείται αυτός ο στόχος του 20%. Δεύτερο σχόλιο, δεύτερο, δεύτερη παρατήρηση. Παράγραφος 37. Όσον αφορά την ερεσιμότητα των ε, στόχων για την αναπτυξιακή βοήθεια. Τι εμπίπτει και τι δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Σήμερα ξέρουμε ότι το σύνολο της εξωτερικής δράσης, δηλαδή του κεφαλαίου 4, και που ουσιαστικά αφορά το 80% των κονδυλίων που αφορούν την εξωτερική δράση, Αυτά όλα τα ποσά θα πρέπει να εμπίπτουν στο στόχο της αναπτυξιακής βοήθειας. Και αυτό επίσης, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, τηρείται αυτός ο στόχος, αυτό το ποσοστό. Η μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν αυτών των εξωτερικών κονδυλίων που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό αφορούν την αναπτυξιακή βοήθεια. Στην παράγραφο 37 γίνεται μια διάκριση από τη μία η βοήθεια και από την άλλη τα υπόλοιπα κονδύλια. Όμως, η σχέση που έχουμε με κάποιες περιφέρειες και με κάποιες χώρες μας οδηγούν στο να έχουμε μία δράση πολλές φορές για στόχους που δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να γίνεται πάντα η διάκριση μεταξύ της αναπτυξιακής βοήθειας και της μη αναπτυξιακής βοήθειας. Πάντως η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των κονδυλίων είναι κονδύλια που αφορούν την αναπτυξιακή βοήθεια, το 80%. Και αυτό το 0,7% για το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 0,2% για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες τηρείται. Και ένα τρίτο σχόλιο που αφορά την παράγραφο 41 του σχεδίου της έκθεσης όσον αφορά την προετοιμασία για την νομοθετική εργασία σίγουρα πρέπει να ομαδοποιηθούν και να συγκεντρωθούν κάποια από τα εργαλεία και τα μέσα. Είναι περίπλοκο το σύστημα χρηματοδότησης και αυτό σίγουρα είναι ένα εμπόδιο για την πιο αποτελεσματική εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννοείται λοιπόν ότι πρέπει να γίνει ομαδοποίηση, ότι πρέπει να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα εργαλεία, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εμποδίζει τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, εάν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, σίγουρα θα ενδυναμωθούν ταυτόχρονα και οι αρμοδιότητες ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στο νέο πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο, οι αρμοδιότητε ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι ενισχυμένε. Τέλος, ένα προσωπικό σχόλιο, συμφωνώ με την Πρόεδρο και στα όσα είπε για την ανάγκη να είμαστε λίγο πιο ρηψοκίνδυνοι, πιο τολμηροί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον είναι παρούσα σε χώρες ε, αναπτυσσόμενες ε, σε χώρες με ιδιαίτερες δυσκολίες και σίγουρα θα πρέπει να δούμε πώς η δράση μας θα γίνει πιο αποτελεσματική, πώς θα γίνει η δράση μας ε, πιο προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες των χωρών αυτών και σίγουρα η ανάληψη κινδύνου είναι απαραίτητη σε αυτές τις πολύ ευαίσθητες χώρες για να είμαστε αποτελεσματικοί. Αλλιώς θα χάσουμε σημαντικές ευκαιρίες και δεν θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε όσο θέλουμε στις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ίσως ναι, αυτό το θέμα του ελέγχου πρέπει να το σκεφτούμε και να το λύσουμε στο μέλλον. Έχω τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ που επίσης θέλει να πει ορισμένα πράγματα, ο Κιμ Έλινγκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ, σύντομα, πάρα πολύ σύντομος, πολύ λίγο έχω να προσθέσω σε σχέση με το συνάδελφο. Όσον αφορά την παρατήρηση και την έκθεση για την ανθρωπιστική βοήθεια, τη βρίσκουμε πάρα πολύ χρήσιμη. Συμφωνούμε με, τον, ε, με τη συλλογική αξιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο το μέσο αναπτυξιακή συνεργασία λειτουργήσε ειδικότερα και με το πόρισμα ότι το μέσο αυτό εξακολουθεί να είναι κατάλληλο για το στόχο που προσπαθεί να επιτύχει. Συμφωνούμε. Επίση, συμφωνούμε και με την έντονη έκκληση στην έκθεση και το σχέδιο ψηφίσματο για ένα ξεχωριστό μέσο ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό το θεωρώ δικαιολογημένο και επίση συμφωνούμε συμφωνούμε ε, βεβαίως με τα σχόλια του κυρίου Γκερέρο Σαλόμ ε, και σήμερα για την ανάγκη συνέχισης ε, της χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας και ειδικότερα του αποθέματος, ε, του αποθεματικού επίγουσας ανάγκης. Όσον αφορά τώρα τη σχέση κόστους ε, και αποτελεσματικότητας, ε, αυτό συνάδει μεγάλο βαθμό που είπατε με αυτό που αποφασίστηκε στην Κωνσταντινούπολη. Προσπαθώ να μειώσουμε το, κάσ, το κόστος των συναλλαγών σε ένα πολυετές πλαίσιο. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό. Να προσθέσω κάτι ακόμη σε σχέση με αυτό που είπε ο συνάδελφος από την ΤΕΦΚΟ, την ανάγκη παρέμβασης σε ευάλωτο περιβάλλον. Το έχουμε κάνει εδώ και πολλά, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά πρέπει να προσέξουμε την ανάγκη λογοδοσίας και την ανάγκη της ε, ευέλικτης παρέμβασης. Αυτά δύο πρέπει να τα εξισορροπήσουμε πρέπει να συμμετέχουμε σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Ερυθρού Σταυρού και μέσω του ΟΗΕ. Παράλληλα θέλουμε να προχωρήσουμε προς το στόχο διοχέτευσης περισσότερης χρηματοδότησης σε τοπικό επίπεδο και είναι κάτι επί του οποίου εργάζομαι και εγώ στο δικό μου επίπεδο. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή αυτή, ε, η συμβολή στη συζήτηση για το επόμενο ΠΔΠ. Δεν ξέρω αν η ΕΕΔ είναι εδώ ή αν θέλει κάτι να προσθέσει. Δεν είναι υποχρέωση. Σας ευχαριστώ. Αν δεν θέλετε να πείτε τίποτε άλλο, να δώσω πάλι το λόγο στον Ενρίκε. Ναι, ευχαριστώ. Ναι. Πρέπει να είναι ε, ο διάλογος στη βάση αυτόν πρότειναν όλοι και ευχαριστώ για τις προτάσεις σας και θα δω πως όλα αυτά θα τα καλύψω, τα λάβω υπόψη όσα είπατε είπατε πολλά για διαφορετικά πράγματα. Α, Φερρυπίν, συμφωνώ με τον κύριο Αγγέλ. Το σύστημα της ενίσχυσης μέσω του προϋπολογισμού budget support είναι περίπλοκο σύστημα. Γιατί έχει χώρες όπου αποδίδει. Αλλά υπάρχουν και χώρες όπου το σύστημα δεν αποδίδει. Τελικά, το πρόβλημα είναι ότι οι χώρες τις οποίες το σύστημα αποδίδει έχουν τις συνθήκες. Οπότε μπορούν να γίνουν τα έργα χωρίς την δημοσιονομική στήριξη γιατί η κυβέρνηση της χώρας έχει τη δυνατότητα και τη βούληση και θέλει και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου. Εκεί που δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα είναι ακριβώς γιατί η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις δεν έχουν αντίστοιχε δυνατότητες. Οπότε και υπάρχουν οι κίνδυνοι του να πάνε τα χρήματα σε άλλες προτεραιότητες. Ή να μην πάνε σε προτεραιότητες και να πάνε σε άλλα, ανομολόγητα. Οπότε θα πρέπει τελικά να βρούμε την ισορροπία και στην περίπτωση όπου μετρημένα θα χρησιμοποιήσουμε την δημοσιονομική στήριξη, να έχουμε έναν μηχανισμό ελέγχου που να είναι πιο στεγανός, πιο αυστηρός και όταν εκχωρηθεί η σχετική υποστήριξη να μην παραλύει ο έλεγχος. Το είπε και ο Φρανκ, το είπε και η Πρόεδρος και όλοι συμφωνούμε. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν επίσης ανομολόγητα συμφέροντα και όχι ξεκάθαρα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση που δρούν εκεί όπου και εμείς παρεμβαίνουμε. Και εκείνοι διέπονται από πολύ λιγότερους περιορισμούς και ελέγχους και άρα μπορούν καλύτερα να ικανοποιήσουν τα όσα ζητούν οι κυβερνήσεις ή ο κόσμος στις χώρες εκείνες. Και όχι επειδή λύνει το πρόβλημα με μια συγκεκριμένη επένδυση, κάτι το οποίο είναι κρυστάλλινο και που άμεσα καλύπτει την καθημερινότητα του κόσμου. Και ό,τι κάνουν, το κάνουν υπονομεύοντας είτε τα, την οικονομική συγκυρία, είτε την πολιτική, για να μπορούν να φέρουν εις το έργο που ανέλαβαν. Και όχι μόνο σε αυτή την έκθεση, αλλά και στο πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον η αναπτυξιακή συνεργασία θα πρέπει αυτή η σκέψη να ληφθεί υπόψη για να μπορούμε όσο γίνεται να είμαστε αποτελεσματικοί. Όσο αποτελεσματικοί και άλλοι στην παγκόσμια σκηνή. Και έτσι με την αποτελεσματικότητα να μπορούμε να αναδείξουμε, να προβάλλουμε αυτές τις αξίες που δεν τις έχουν οι άλλοι. Τώρα, σε σχέση με τα όσα είπε που έφυγε. Ε, βέβαια συμφωνώ, είναι βασική υπόθεση για την ε, Επιτροπή μας, το να αποκτήσει ανθεκτικότητα και αντοχή αυτή μας η πολιτική, να μπορούμε να προσδώσουμε σε αυτές τις κοινωνίες κάποιες δυνατότητες, οπότε από μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Και στην οικονομική πολιτική και σε άλλες πολιτικές, στην παιδεία, στην υγεία, σε ό,τι μας απασχολεί. Είναι θέμα διακυβέρνησης, όλο είναι και πιο σημαντικό για τους διάφορους μηχανισμούς που παρέχουν σε αυτές τις δυνατότητα να μπορούν ε, από τη δομή των θεσμικών του οργάνων να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Και εδώ κολλάει αυτό που είπε η Μαρία. Δηλαδή ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό για την ε, ειρήνη και τις πολιτικές, για διακυβέρνηση, χρηστή διακυβέρνηση που διαβόνται από τις γνωστές αξίες μας. Για την Επιτροπή τώρα. Πήγαμε στο 20% για κοινωνικές υπηρεσίες και παιδεία. Καλά μαντάτα είναι αυτά και δεν μπορούμε παρά να χαρούμε γι' αυτό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε το 20% όπως προβλεπόταν από τον αντίστοιχο μηχανισμό όταν αυτός συγκροτήθηκε. Ε, λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα τα της παραγράφου 37 για τον 90%. Θα πρέπει να βρεθεί κατάλληλη διατύπωση ότι δηλαδή έχουμε εδώ πέρα για εξαιρετικούς λόγους και γι' αυτό συγκεράζουμε, αναμειγνύουμε διαφορετικές δράσεις, ψυχική βοήθεια και άλλους μηχανισμούς, οπότε τουλάχιστον να μπορούμε να πετύχουμε διαφάνεια, να πετύχουμε λογοδοσία και ιδιαίτερη προσπάθεια Δηλαδή κάτι, να, να, να φτιάξουμε κάτι που δεν είναι ε, αναπτυξιακό, να το, να το φτιάξουμε, να το, να το ε, μασκαρέψουμε τέλο πάντων να μοιάζει με ανάπτυξη, να το φτιασιδώσουμε. Και αυτό είναι σημαντικό που βέβαια όμως εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας άπαξ και αποδίδουν κάποιοι μηχανισμοί. Αυτό γίνεται γιατί η Κομισιόν παρουσιάζει μια γενική ρότα για όλες τις πολιτικές αυτών των μηχανισμών, όχι μόνο για τις πολιτικές εξωτερικής δράσης ή μόνο για τις πολιτικές ε, ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας. Οπότε και θα ακολουθήσει συζήτηση και διαπραγματεύσεις και αναμέτρηση ενδεχομένως μεταξύ Κομισιών Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Μάλλον αυτό θα βρούμε μπροστά μας τους αμέσως επόμενους μήνες. Και επίσης, ευχαριστώντας τον Επίτροπο της Κομισιόν που είχε την καλοσύνη να έρθει να τα πούμε για να ετοιμάσω αυτό το κείμενο, θέλω λίγο να του πω ότι κατόπιν της συνάντησή μας εγώ πήγα σε μια ακρόαση στην ΑΦΕΤ που του, ταυτόχρονα ετοιμάζει μια έκθεση για τους μηχανισμούς εξωτερικής δράσης και αυτό το οποίο απεκόμισαν ότι το Κοινοβούλιο γενικότερα και μόνο η Επιτροπή μας προσπαθεί και, και κατατείνει προς μια ενοποίηση. Και αυτό όμως γίνεται με κάποιο είδους γενικότερη συνένεση. Βέβαια ο καθένας θέλει το δικό του και έχουμε πάρα πολλές φήμες, φήμες και όχι πληροφορίες ότι ακόμα και στην, ε, ε, στην υπηρεσία της Επιτροπής για την Εξωτερική Δράση ούτε εκεί υπάρχει ομοφωνία. Για να δούμε τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Τέλος πάντων, επιμένω το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι αυτό το θέμα δεν ε, είναι δικής μας μόνο αρμοδιότητας και αν ε, δρομολογηθούν κάποιες εξελίξεις αυτό θα οφείλεται σε μια γενικότερη πρόταση της Κομισιόν που θα υπόκειται σε έγκριση όλου του Κοινοβουλίου μέσα από διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο που <laughs> μοιραία θα έχει επιφυλάξει κάποιο είδους. Ο εκπρόσωπος της ΕΚΟ. Ξέρουμε εδώ στην Επιτροπή μας ότι είμαστε εναφανδόν υπέρ της ανθρωπιστικής δράσης της Κομισιόν. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι κανείς να καλύψει κρίσεις που πολλές φορές είναι προσδόκητες, που χρειάζονται από βιαιότητα. Και πολλές φορές φύγουν εκατομμύρια. Α, η Συρία τώρα μπήκε σε κάποια ομαλότητα αλλά τώρα ξέσπασε άλλη κρίση που πρόκειται επίσης να θίξει εκατομμύρια. Τα ερήπια και άλλη κρίση που επίσης χαρακτηρίζεται από ένταση και βία. Οπότε χρειάζεται η πιο μεγάλη ευελιξία για να μπορέσει κανείς να βοηθήσει να βοηθήσει ε, πάρα πολύ σε καταστάσεις που απαιτούν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Και με τη Λίντα σύμφωνα, Πολλές φορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι και η πιο ευέλικτη ε, από όλες τις, ε, τις διεθνείς πλατφόρμες ε, έχει ακριβώς αυτή την ε, έλλειψη ευελιξίας που εμποδίζει, εμποδίζει την ε, δημιουργικότητα και έτσι φρενάρεται κάτι που χρειάζεται κάποιο τομέας, κάποιο μέρος και πολλές φορές πολλά από αυτά τα προβλήματα θα λυνόντουσαν με έναν πιο εντατικό διάλογο, με περισσότερη αμοιβαία εμπιστοσύνη, φερειπίν μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου θα μπορούσε να προτείνει η Κομισιόν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ε, να έχουν καινοτόμο χαρακτήρα πέραν του ρυθμιστικού πλαισίου και να θεωρήσουμε ότι αξίζει αυτή η κοινοτομία και έτσι να βγει μια συμφωνία σημαντική ουσιαστική. Ευχαριστώ πολύ, Ενρίκε. Πριν σας δώσω την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, θα ήθελα να πω ότι ότι ο Χουάν Κάρλος εδώ μας βοήθησε πάρα πολύ και είναι η τελευταία επιτροπή ε, στην οποία συμμετέχει. Θα φύγει γιατί είμαστε και πάλι θύμα της κινητικότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φεύγει ο Χουάν Κάρλος από εμά και πάει στο Eurolat. Δουλεύει για μας εδώ και 7 χρόνια, έχει πάρα πολύ εμπειρογνωμοσύνη, την οποία ε, συνεισέφερε στην Επιτροπή μας, ειδικότερα στο κομμάτι της ανάπτυξης. Θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω τις ε, ευχαριστίες μας ε, ε, στον Χουαν Κάρλος. Ελπίζουμε να το δούμε στο Eurolat με την οποία συνεργαζόμαστε. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για όλα όσα έκανες για την Επιτροπή μας, Χουαν Κάρλος. Και καλή συνέχεια. Ο Ενρίκε θέλει κάτι να πει. Εγώ θα τον ευχαριστούσα όταν κλείσει και εγκριθεί η έκθεση. Κανείς δεν ξέρει πού θα πάει η υπόθεση και πού θα καταλήξει η έκθεση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όμως πρέπει να σας πω ότι εντάξει δεν έγινε τίποτα για αυτή την έκθεση πλευρά του Χουάν Κάρλος. Θα μπορούσε να ε, ε, ονομάζεται Ερέρο Χουάν Κάρλος η, έκθεση. Α, ωραία, τότε να το θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ευχαριστίε από πλευρά του Ενρίκε το πόσο σε βοήθησε και για αυτή την έκθεση έχουμε 27 Φεβρουαρίου το μεσημέρι ε, τροπολογίες και 23 η ψήφιση. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο προχωρούμε. Item, which is also an που είναι επίση πολύ σημαντικό, το οποίο κάπως το συζητήσαμε προηγουμένως και με τον κύριο Στάινερ, το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρεί τι προϋποθέσεις, συγγνώμη, τις δεσμεύσεις της του 0,7% ε, ε, του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματος πριν από τρία χρόνια αποφασίστηκε η αλλαγή του συστήματος και να μην δημοσιεύεται αυτή η έκθεση λογοδοσίας, ε, τότε έτσι την αποκαλούσαμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έλεγε ότι δεν το έκανε πια γιατί προσπαθούσε να προσαρμοστεί και θα κάνει υποβολή εκθέσεων για τους ε, ε, στόχους αηφόρου ανάπτυξης. Ε, κάποιοι είπαν ότι επειδή δεν καταφέρνουμε το 0,7% δεν θέλαμε ακριβώς να επικεντρώνεται η προσοχή σε αυτό. Μετά από το 2005, από όταν, κάναμε, όταν ε, ε, αναλάβαμε τις πρώτες δεσμεύσεις, πάρα πολλά κράτη-μέλη δεν φτάνουν στο 0,7%. Η ε, συνάδελφος Χόιμπορκ από, το, από, τους Πράσινους ζήτησε να γίνει αυτή η συζήτηση εδώ και θέλουμε να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΕΔ Πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με το 0,7% για τι έχει να κάνει και με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, που είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στην Επιτροπή μας. Η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, λοιπόν, Λογόν ε, Σάριζεν, είναι εδώ μαζί μας ε, και βέβαια μετά θα λάβει το λόγο και η ΑΕΔ. E Κύριε Σάριζεν, έχετε το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Sorry. Uh, yes, I do have water. Thank you. Έχω νερό. Ευχαριστώ. So indeed we had this Ναι, πράγματι, για τρία χρόνια είχαμε σταματήσει αυτή την έκθεση λογοδοσίας, όπως την αποκαλούσαμε και όπως είχε προγραμματιστεί και είχε ανακοινωθεί θα ξαναρχίσουμε την ε, ε, υποβολή νέας έκθεσης που τη λέμε χρηματοδότηση ε, για την αναπτυξιακή βοήθεια. Έχουμε σκοπό να το δημοσιεύσουμε για την χρηματοδότηση του Φόρουμ της Ανάπτυξης που θα λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη στις 23 με 26 Απριλίου. Οπότε έχουμε ένα πρώτο σχέδιο της έκθεσης, ε, ε, για την ώρα ένα, πρώτο, ένα προσχέδιο της έκθεσης, αλλά δεν ε, απέχει πολύ ακόμη από την ολοκλήρωσή του. Βέβαια, τα προσωρινά στοιχεία της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας γίνονται, δημοσιεύονται και είναι επίσημα μέσα Απριλίου. Για την ώρα δεν έχουμε καμία απολύτως ένδειξη ποια θα είναι τα στοιχεία αυτά για το 2017. Ο στόχος ε, της νέας έκθεσης ε, είναι να γίνει μια υποβολή εκθέσεων για τους διάφορους τομείς δραστηριότητας ε, της, του θεματολογίου που καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη, τα κεφάλαια βασίζονται στα βασικά θέματα της ε, Ευρωπαϊκής Συνένεσης. Και ένα σημαντικό σημείο ε, στο οποίο επικεντρωθήκαμε είναι να δούμε και τα χρηματοδοτικά και τα μη χρηματοδοτικά μέσα εφαρμογή, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι ε, όλο το νόημα του θεματολογίου αυτού, να υπάρχει δηλαδή συνδυασμό των χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών πτυχών, θα πρέπει να καλύπτονται όχι μόνο, ε, θα πρέπει να καλύπτονται και αυτά στην έκθεση, όχι μόνο η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, η οποία θα παραμείνει ένα σημαντικό τμήμα τη έκθεσης, αλλά η έκθεση θα εξετάσει όλες τις δεσμεύσεις ε, την ε, ε, της, ε, του θεματολογίου της Αντίσα ε, Μπέμπα. Υπάρχουν, υπάρχει κινητοποίηση των ε, εγχωρίων πόρων, η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία, το διεθνές εμπόριο ως κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης, ζητήματα υφορίας, επιστήμη, τεχνολογία, καινοτομία, δεδομένα παρακολούθησης και ελέγχων. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν ε, για όλα αυτά τα θέματα θα συνδυαστούν με μια αξιολόγηση της επίδοσης και ε, των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών μελών για όλους αυτούς τους τομείς. Όπως είπα, ε, θα επικεντρωθούμε επίσης και ε, στα βασικά σημεία εστίασης της Ευρωπαϊκής Συνένεσης. Η έκθεση θα εγκριθεί ως ε, έγγραφο εργασίας του προσωπικού, ελπίζουμε πριν από το φόρουμ. Είναι βέβαια πολύ δύσκολο το χρονοδιάγραμμα, γιατί ένα μήνα πριν θα γίνει ε, το φόρουμ από ό,τι γινόταν μέχρι τον περασμένο χρόνο. we do hope to Ελπίζουμε όμως να τα καταφέρουμε. Όσον αφορά την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, ε, θα έχετε δει τα τελικά στοιχεία για το 2016, τα οποία δημοσιεύτηκαν το Δεκέμβριο και θα είδατε ότι η, τα στοιχεία για το 2016 είναι 77,7 δις ε, ευρώ, ε, δηλαδή δεν επιτυγχάνουμε ακόμη το 0,7 της 100. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως ευχαρίστως να σημειώσουμε ότι υπάρχει μία πρόοδος ε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα και ειδικά ειδικότερα ως προς τη βοήθεια προς τις χώρες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία, ένα από τα βασικά μηνύματα της επερχόμενης έκθεσης σε σχέση με την επίσημη αναπτυξική βοήθεια στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ε, για τις οποίες ε, ε, απέχουμε πολύ από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων. For Για τα υπόλοιπα, η έκθεση θα συμπεριλάβει δείκτες για κάθε ε, υποχρέωση, για κάθε ε, πίστοση. Θα υπάρχει μία γραφική παράσταση που θα δείχνει πού βρίσκεται συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και από απόψεως προσπάθειας και από προσπάθειας αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί για τις ε, διάφορες ε, υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ε, στην Αντισαμπέμπα. Είναι πολύ νωρίς να σας δώσω πάρα πολλές λεπτομέρειες για τους δείκτες αυτούς, γιατί όπως είπα ακόμη καταρτίζουμε την έκθεση και επειδή συμπεριλαμβάνει έκθεση πληροφορίες ε, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τα κράτη-μέλη, για κάποιους δείκτες ακόμη είναι λίγο δύσκολο να δούμε πού βρισκόμαστε γιατί κάποια κράτη-μέλη ε, αναφέρονται πολύ, κάποια άλλα πολύ λιγότερο, οπότε η εικόνα δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκιαγραφηθεί. Όμως ελπίζουμε ότι θα το επεξεργαστούμε και θα είμαστε έτοιμοι να το παρουσιάσουμε στα μέσα του Απριλίου πριν από το ε, φόρουμ EFFD. Ε, και ευχαρίστω να ε, συζητήσουμε την έκθεση αυτή στην ομάδα. Πότε γίνεται αυτό το φόρουμ, 23 με 26 Απριλίου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και πότε θα είναι έτοιμη η έκθεση. Ελπίζουμε για εκείνες τις ημερομηνίες να το έχουμε έτοιμο. Αρχές Απριλίου ελπίζουμε να είναι έτοιμο όμως. Πρέπει να προσθέσουμε τότε τα στοιχεία της ε, επίσημης αναπτυσσικής βοήθειας, τα οποία θα τα λάβουμε από τον ΩΣΑ στα μέσα Απριλίου. Οπότε τσίμα τσίμα, δηλαδή ακριβώς πριν την ημερομηνία. Εντάξει. Καλό θα ήταν να συγκεντρώσουμε όλα τα σχόλια, αυτά που ακούστηκαν στη Νέα Υόρκη, αυτά που είπαν οι άλλοι εταίροι. Το σημειώνουμε. Μαρία, εσύ εσύ έτσι και το έβαλες το θέμα αυτό σε αυτή την ημερήσια διάθεση. Ευχαριστώ πολύ Λίντα. Ευχαριστώ την Επιτροπή. που ανταποκρίθηκε σε αυτή την έκθεση, μας έκανε την παρουσίαση γιατί εμείς ε, δεν ε, προλάβαμε να την συζητήσουμε. Βλέπω ότι ουσιαστικά δημιουργείται εδώ μια εικόνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα κράτη-μέλη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Και το ερώτημα είναι αν προχωράμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Μας είπατε ότι υπάρχει συμφωνία, ότι μέχρι το 2015, ότι μέχρι το 2015 υπήρχε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και ότι ολοκληρώθηκε το 70% του στόχου. Σήμερα όμως έχουμε σχέδιο. Εσείς, σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να ολοκληρωθεί η επίτευξη του στόχου και βεβαίως περιμένουμε με ανυπομονησία την έκθεσή σας και σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχουμε ήδη πάρει και από το να υλοποιηθεί το υπόλοιπο κομμάτι των στόχων. Μας λέτε ότι το 70% έχει ήδη, επαναλαμβάνω, επιτευχθεί και θα αναφερθεί το θέμα αυτό στο πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο. Μπορείτε να μας πείτε ποια ακριβώς αναφορά θα γίνει για το πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο σε σχέση με τους στόχους αυτούς. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε τι νέος κωδικός προβλέπετε για την μετανάστευση, καθότι η Αυστραλία, οι Ηνωμένε Πολιτείες, ο Καναδάς δεν έχουν εκφραστεί κατά της πρωτοβουλίας της Επιτροπής. Παραδείγματος χάρη το blending, το θέμα των εγγύσεων. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό, είτε ε, για το θέμα της ε, επιδότησης ε, αγροτικών προϊόντων, γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε καθόλου σκεφτεί αυτές τις ε, προτάσεις. Τι έχετε να μας πείτε για όλα αυτά. Okay, a lot of questions. I didn't... Πολλές ερωτήσεις. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Όχι. Να απαντήσει όλες αυτές τις πολλές ερωτήσεις Μαρίας, λοιπόν, η Επιτροπή. Thank you. Uh, Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην ξεχάσω όλες αυτές τις ερωτήσεις. Καταρχήν το ποσοστό των ε, στόχων 20% είναι για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και στα πλαίσια της επόμενης αξιολόγησης του πολιετούς θα πρέπει βεβαίως να τεθούν τα νέα ποσά μάλλον ε, θα μειωθεί το ποσοστό της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Δεν έχω καμία τελική, αν θέλετε, σκέψη. Αλλά αυτό το 0,7 πιστεύω ότι είναι κάτι που θα το διατηρήσουμε. Τώρα, όσον αφορά τις δημιουργίες των κρατών μελών και τον τρόπο να τις στηρίσουν, εμείς πιέζουμε όσο μπορούμε, χρησιμοποιούμε όλες τις ευκαιρίες να τους υπενθυμίσουμε τις δεσμεύσεις τους και ότι αυτό το 0,7% πρέπει να τηρηθεί. Και οι ατομικές δεσμεύσεις αλλά και οι συνολικές δεσμεύσεις ε, είναι κάτι που παρακολουθούμε να τηρούνται. όσον αφορά τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και τα επιμέρους στοιχεία σίγουρα τα δικά μας δεδομένα έχουν αν θέλετε λιγότερη βαρύτητα από αυτά του ΟΣΑ. Τι άλλη πίεση αν θέλετε να ασκήσουμε εμείς. Νομίζω ότι η δημοσίευση των στοιχείων του ΟΣΑ είναι κάτι που συζητείται σε αιτήσια βάση από το Συμβούλιο και υπάρχει αναφορά αυτών στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και φυσικά αυτό έχει αρκετή βαρύτητα πιστεύω και ασκεί αρκετή πίεση προς τα κράτη-μέλη. Το θέμα του κωδικού This is not meant... το θέμα του κώδικα για τη μετανάστευση δεν θέλουμε εδώ να επεκτείνουμε και να διευρύνουμε το εύρος των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. όσον αφορά τη μετανάστευση συμπεριλαμβάνεται ναι ή όχι στους στόχους. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να σας το απαντήσω με βεβαιότητα. Ε, Uh, το θέμα του κωδικού για την μετανάστευση του DAC είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει και δεν έχουμε πρόθεση να διευρύνουμε καταρχήν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε άλλους τομείς που δεν καλύπτονται σήμερα από την παρούσα ε, χρηματοδότηση. Θέλουμε να συμπεριλάβουμε και εργαλεία του ιδιωτικού τομέα και σίγουρα έχουμε επεξεργαστεί εδώ και αρκετό καιρό τους κανόνες για το θέμα του blending και στο δημόσιο τομέα, όχι ακόμα στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει συμφωνία ως προς τον ιδιωτικό τομέα ακόμα. Θέλουμε να βρεθεί μία αντιστοιχία προς το blending, και βεβαίως όταν αποπληρώνονται τα δάνεια υπολογίζεται στους ε, στόχους και τα περισσότερα μέλη του ΝΤΑΚ θεωρούν ότι υπάρχουν στοιχεία αυτών των ε, δανείων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν ε, σε αυτό το blending. για την ε, επιδότηση των ε, αγροτικών προϊόντων, γιατί κάνατε και αυτή την ερώτηση. Αυτό όχι δεν προβλέπεται να συμπεριληφθεί. Και εδώ συζητείτε τα πλαίσια του PSI και άλλου είδους χρηματοδότησης που συνυπολογίζεται. Παραδείγματος χάρη είναι επιδότηση ε, και εγγύηση εξαγωγών σε αυτά τα πλαίσια. Η Έλλη. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά καθυστέρησα. Σήμερα υπάρχουν πολλές ε, επιτροπές που συνεδριάζουν. Ξέρω ότι η Χάιντι, συνάδελφός μας, έχει υπενθυμίσει ήδη ότι την τελευταία φορά που συνεδρίασε η ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη και τη μετανάστευση συζητήθηκαν αυτά τα θέματα και εκφράστηκαν και κάποιες ανησυχίες. Όπως είπατε, δεν υπάρχει σαφής πρόθεση να διευρυνθεί η αιρεσιμότητα, να προσθεθούν και άλλοι, άλλες δυνατότητες. Αλλά όλοι θέλουμε νομίζω να υπάρξει μια μεγαλύτερη σαφήνεια για τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση θεμάτων που άπτονται της μετανάστευσης. Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που βρίσκονται λίγο στο μετέχμιο. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να τις θεωρήσει σαν ε, προγράμματα ή δραστηριότητες καθαρά αναπτυξιακές. Και η ανησυχία μας είναι ότι αν προσθεθούν νέα κριτήρια και δεν επιτρέψουν κάποιες δαπάνες να καταχωρηθούν σε αυτούς τους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης ή δεν καταχωρηθούν σαν αναπτυξιακή βοήθεια στους παραδοσιακούς τομείς αναπτυξιακής βοήθειας, όταν μιλάμε παραδείγματος χάρη για δάνεια για άλλου είδους βοήθεια, τη λεγόμενη tight aid, χρειαζόμαστε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Τα προηγούμενα χρόνια είδαμε ότι αυξήθηκαν οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς ασφάλειας, άμυνας τα τελευταία δέκα χρόνια. Κινδυνεύουμε λοιπόν να δούμε όλο και περισσότερα ποσά να μην έχουν ε, χαρακτηρισμό καθαρά αναπτυξιακό, γιατί βρίσκονται στο μετέχμιο κάποιων δραστηριοτήτων που είναι όχι μόνο αναπτυξιακές ή αναπτυξιακές και κάτι άλλο. Και αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να το προσέξουμε. Αυτό που ονομάζουμε λοιπόν ε, επαυξημένη βοήθεια, inflated aid, θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το 0,7% και η επόμενη περίοδος, δηλαδή μέχρι το 2030, γιατί οι πρώτοι στόχοι ουσιαστικά τέθηκαν για το 2015 πριν από μισό αιώνα. Στις επόμενες λοιπόν προσφορές των δωρητών στις επόμενες ε, συνεδριάσεις για υποσχέσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να δούμε πώς θα διατηρήσουμε τα ποσά αυτά και τα επίπεδα χρηματοδότησης. Βλέπουμε στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ότι τα ποσά τα οποία απευθύνονται σε αυτές μειώνονται διαρκώς. Και κάποια ταμεία όπως το Trans Fund for Africa το οποίο οι δαπάνες απευθύνονται σε μεγάλο βαθμό σε χώρες ε, που βρίσκονται κοντά στην Ευρώπη ή στις διαδρομές αυτών που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Και η ανησυχία μας είναι ότι άλλες χώρες εγκαταλείπονται, τις ξεχνάμε, τις χρηματοδοτούμε όλο και λιγότερο. Όπως είπε ο κύριος Στάινερ νωρίτερα, αν δεν παίξει καθοριστικό και ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, ποιος άλλος θα το κάνει. Ποιος άλλος θα παίξει αυτό το ρόλο. Γιατί βλέπουμε ότι άλλοι μεγάλοι παίκτες της αναπτυξιακής βοήθειας εγκαταλείπουν το πεδίο και το ρόλο τους. Η Μαρία. Δεν θέλω να επανέλθω, γιατί δεν συμφωνώ με την απάντησή σας όσον αφορά αυτό που είπατε για τις επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων. Όταν λέτε ότι ο νέος κωδικός DAC για τη μετανάστευση είναι μόνο για θέματα διαφάνειας. Εδώ βλέπουμε καθαρά ότι για την μη εθελοντική επιστροφή υπάρχουν κάποια ποσά και κάποιες δαπάνες που καταχωρούνται και εδώ αυτός ο νέος ε, κωδικός για τη μετανάστευση θα συμπεριλαμβάνει ενδεχομένω και αυτά τα ποσά. Δεν είναι μόνο θέμα διαφάνειας αν θέλετε και αναρωτιέμαι πραγματικά αν ε, συμφωνείτε ότι πρέπει να υπάρξει ένα μείγμα μέτρων, ένα μείγμα πρωτοβουλειών. Και βεβαίως μπορεί κανείς να προσθέσει και άλλες δραστηριότητες και άλλες πρωτοβουλίες και να αυξηθεί ο κατάλογος. Αλλά δεν συμφωνώ απολύτως με την απάντηση που δώσατε για το θέμα αυτό. Σε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει σε κάποια από αυτά γιατί μερικά τα καλύψατε με την παρουσίασή σας. Ε, Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια παρεξήγηση όσον αφορά το τι προτείνουμε για αυτό τον κώδικα, κωδικό. για την μετεγκατάσταση γιατί εν προκειμένου με τη μετακατάσταση θα υπάρξει μετακίνηση. Θα πάνε οι πρόσφυγες από τις αναπτυσσόμενες χώρες σε άλλες αναπτυσσόμενες ή στη δική τους χώρα, όπου υπάρχει η βούληση προς τούτο. Έτσι προβλέπεται τώρα και εμείς δεν θέλουμε να τα αλλάξουμε. Πρόκειται μόνο περί εθελουσίας επιστροφής. Δεν έχουμε πρόθεση μεταβολής του καθεστώτος. από τις δικές μας χώρες σε άλλοι αναπτυσσόμενοι στη δική τους. Για τα άλλα τώρα. όσον αφορά τον ορισμό της επίσημης ανησυχικής βοήθειας. και της Titan θέλουν η, η ενίσχυση αυτή να μην καλύπτεται από την ODA. Η μη αυξημένη βοήθεια δηλαδή. Και είναι θέμα αποτελεσματικότητας. Τέλος πάντων αποτελεσματική όχι παραμένει μια ενίσχυση. Επομένως παραμένει και η Tide μια τέτοια ODA επομένως προσπαθούν οι χώρες να αυξήσουν την προσφερόμενη κάλυψη και τον δανεισμό μας στον τον Μα Αυτό είναι και το ζουμί του θεματολογίου της Αντισαμπέμπα. Το πώς θα βοηθούν τις όμορες χώρες, δηλαδή το πώς θα μπορούμε να αντιλήσουμε πόρους και το ODA είναι ο καταλήτης για να συγκεντρώσει κανείς αυτούς τους έξτρα άλλους πόρους Άρα να δημιουργήσουμε το κίνητρο ούτως ώστε οι δανειστέ να δώσουν και άλλα οι δωρητές τέλος πάντων. Και οι άλλοι πόροι που θα ελκυστούν είναι ο ιδιωτικό τομέα. Και έτσι να υπάρξει ισοδύναμο δανείο. Τώρα, όσον αφορά τι δαπάνε για του πρόσφυγε. ε, αυτό καλύπτεται εδώ για πολλά χρόνια από τα ODA. Και η πρώτη αύξηση των ε, προσφύγων προς την Ευρώπη οδήγησε και στην αύξηση του ODA. Από το 16 δηλαδή και μετά οι δαπάνες ανήλθαν στο 25% περίπου της αυξήσεως του ODA για το σύνολο της ενώσεως. Since the, uh, <coughs> the movement of refugees have, have και οι ροές των προσφύγων το επιτοπλίστων όμως τώρα έχουν φρενάρει και επομένω. Αυτέ οι δαπάνε των δωρητών ε, μόνο για ένα χρόνο μηχανικά καλύπτονται για το 17. Οπότε περιμένουμε να μας πούν τα στοιχεία για αυτή τη χρονιά γιατί μετά υπάρχει μείωση παρά το ότι συνεχίζουν και καταβάλλονται δαπάνε φιλοξενίας των προσφύγων παρά το ότι πλέον δεν επιλέξουμε σε δαπάνε για όντιο, επομένω. Περιμένουμε τώρα να μάθουμε ποια είναι τα στοιχεία. Περιμένουμε όμως τι θα γίνει για τη χρήση του 17, πού έχουν φτάσει τα σχετικά νούμερα. Για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ODA, το είπαμε στην αρχή, μα για αυτό είπαμε ότι ανησυχούμε, γιατί απέχει πολύ από το να τηρήσει τα υπεσχημένα η Ευρωπαϊκή Ένωση. ODA για τις LDCs, τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Μακάβαν. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι έχετε καλή. Α, η Έλλη, Έλλη. Α, γιατί Έλλη, πες τα γρήγορα, γιατί άργησε, αλλά ήρθε ο Σάρλ. Πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Είπατε επίση ότι δεν τίθεται σε συζήτηση πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί απλώ αμφισβητούμε την ιδέα ότι σε κόστο ε, προσφύγων, ε, προσφύγων ε, σε δολάρια, αυτές είναι οι, αυτά είναι τα πόσα, γιατί μιλήσατε για κάποια ομαδοποιημένα στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά για κάποιε χώρε όπω η δική μου, η Ιταλία για παράδειγμα, πηγαίνει προς πολύ κακή κατεύθυνση και ανεξέλεγκτα Είμαστε στο 0,26 αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, αλλά να αφήσουμε το κόστος, ε, τα ποσά για τους πρόσφυγες είναι ακόμη λιγότερα. Ε, σε μερικές χώρες ε, λοιπόν υπάρχει τεράστια διαφορά και απόκληση από το στόχο. Νομίζουμε ότι αυτό δεν είναι δίκαιο και γι' αυτό ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε αυστηρότερα κριτήρια, τουλάχιστον για την επαλήθευση του κατά, του πόσο είναι... ε, ε, γνήσια τα αποτελέσματα αυτά που προσμετρώνται ως αποτελέσματα από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Όμως δεν είναι κανόνες αυτές Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει η Πρόεδρος. Αυτά είναι ε, κανόνες DAC. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τις αποφάσεις, αλλά δεν αποφασίζουν εκείνοι. Σαρλ, άργησες. Ε, αν είσαι σύντομο όμω, μπορεί να θέσει και εσύ τα ερωτήματά σου. Ναι, πάρα πολύ γρήγορα. Το ζήτημα, της συζήτησης, το ζήτημα της συζήτησής μας τώρα είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαγγέλλεται συνεχώς αλλά ποτέ δεν ε, λαμβάνει χώρα. Πολλές φορές έχει γίνει αυτό στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί για να ε, κινητοποιήσει τα κράτη-μέλη για να προοδεύσουν, όμως ε, δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα έπρεπε να είναι εδώ, αλλά τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα έπρεπε να μας πούν για ποιο λόγο δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο στόχο. Τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να μας πούν αν ναι ή όχι έχουν κάνει υποσχέσεις. Έχουν κάνει υποσχέσεις, το ξέρουμε αυτό του 0,7% εδώ και δύο χρόνια πριν από την Αντίσα Μπέμπα ε, το είχαν κάνει πριν από 15 χρόνια το λοιπόν που βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ένα ε, κημητήριο των υποσχέσεων, είναι ένα κέντρο ανακύκλωσης υποσχέσεων για να το πω έτσι. Γίνονται υποσχέσεις, δεν τις ε, σεβόμαστε και τις ξανακάνουμε. Το κάναμε το 2000, το κάναμε το 2015, κάθε φορά με έναν ε, ορίζοντα 15 ετών, το ξανακάνουμε το 2030. Το είχαμε ξαναπεί στην Επιτροπή αυτή, ότι τα κράτη-μέλη που έχουν υποσχεθεί κάτι τέτοιο πριν από την Αντισαμπέμπα, που ήταν στο 0,4%, που δεν έκαναν τίποτα από τότε, δεν θα φτάσουν ποτέ να φτάσουν στο 0,7% το 2030. Γιατί θα έπρεπε να αυξήσουν ε, την αναπτυξιακή βοήθεια τους, ε, ε, την αναπτυξιακή βοήθεια του κατά 0,02% κάθε έτος. Αν το κάνουμε αυτό γραμμικά δεν πρόκειται να συμβεί. Οπότε πρέπει να Πρέπει το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευθυγραμμιστούν, να συντονιστούν για να ε, έχουν μια πιο ισχυρή αντίδραση. Να περιμένουμε τον Απρίλιο, να δούμε πώς θα είναι η έκθεση, θα είναι απογοητευτική σίγουρα. Μέχρι τότε πρέπει να σκεφτούμε μια στρατηγική για να, ε, να μην ε, μας κοροϊδεύουν, να μην μας πιάνουν κορόιδα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει τίποτα άλλο να προσθέσει. Νομίζω ότι η, αυτό που είπε η Έλλη δεν ε, είναι στο χέρι σας. Το πώς δηλαδή αποφασίζονται οι κανόνες DAC ε, είναι κάτι που πρέπει να, για το οποίο πρέπει να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας. Εμείς πρέπει να ασκήσουμε πίεση στις κυβερνήσεις μας. Προκύπτει και από αυτό που είπε ο Σάρλ για το θέμα αυτό. Το να επεκτείνονται συνεχώς τα μέτρα είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ο κύριος Γκέρενς πρέπει να μην ε, είμαστε πια ε, αφελείς, να νομίζουμε ότι θα γίνει και θα φτάσουμε στο 0,7%. Οι μόνοι που το κατάφεραν είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, όλος προσφάτως, γιατί το έγραψαν αυτό σε νόμο. Πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι δεσμευτικό, να μπορεί να υποχρεώνει αυτούς που ανέλαβαν την υπόσχεση, να μπορούν να λογοδοτήσουν και σε εθνικό επίπεδο και εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πράγματι το ε, θα το θέσουμε αυτό και με τους εθνικούς βουλευτές όπως το έχουμε ξανακάνει. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα μετά από την συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη και μπορούμε να συζητήσουμε ε, στους συντονιστές του μηχανισμό για τη διατήρηση της πίεσης από την πλευρά μας. Να περάσουμε στο τελευταίο σημείο για σήμερα, το 22, που είναι η ώρα των ερωτήσεων. Δύο ερωτήσεις έχουμε. Η πρώτη είναι από μένα. Είναι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν, θα σας τη διαβάσω, θα σας πω περί τίνος πρόκειται. Οι Human Rights Watch ε, έχουν καταρτήσει μια έκθεση για την Τανζανία ε, κατόπιν ανακοίνωση του Προέδρου της ε, ότι έγκυες, έγκυες φοιτήτριες, ε, έγκυα, ε, έγκυα, κορίτσια της, δεν μπορούν να συμμετέχουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Απαγορεύεται. αυτό αναφέρεται στην έκθεση της Human, της Human Rights Watch έχει γίνει καμία συζήτηση από πλευρά σας με τις αρχές της Τανζανίας για αυτό το θέμα, γιατί μου φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ άδικο νεαρά κορίτσια επειδή ε, είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης να μην συμμετέχουν στη σχολική εκπαίδευση. Ποιος είναι εδώ, εν πάση περιπτώσει πείτε μας εσείς ποιος είστε ή εσείς ποια είστε. Ε, ευχαριστώ. Καλησπέρα. Μισέλα Μποέν ε, από το κέρας της Αφρικής. Υπεύθυνη για το κέρας Αφρικής. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Γνωρίζει πολύ καλά την έκθεση της Human Rights Watch η Επιτροπή και στάλει μάλιστα 30 Ιανουαρίου στον αρμόδιο επίτυπο Μίτσα. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά όλες αυτές ε, τις ε, αναφορές, ανησυχούμε για την κατάσταση των νεαρών ε, γυναικών και μητέρων και ο ίδιος ο Επίτροπος ε, Νιμίτσα παρακολουθεί το θέμα αυτό με μεγάλη προσοχή. Ο Δόκτωρ Μαρίγκα αλλά και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν επίσης ε, ενημερωθεί και παρακολουθούν το θέμα. Η νέα συμφωνία αναπτυξιακής βοήθειας που υπεγράφει με τον ε, Υπουργό Εξωτερικών της Τανζανίας μας οδήγησε και σε επιπλέον επαφές σε πολύ υψηλό πολιτικό επίπεδο. Οι εκπρόσωποι της χώρας αυτής έχουν επίσης λάβει υπόψη τους τις αναφορές και τις ανησυχίες μας και αυτός διότι έχει αναφερθεί το θέμα αυτό καθώς και η ε, καταναγκαστική γάμη ε, πολύ νεαρών κοριτσιών σε πολλές συνεργασίες, το θέμα των ε, πολύ νεαρών κοριτσιών που αναγκάζονται να παντρευτούν, των νέων κοριτσιών που ε, γίνονται μητέρες, των κακομεταχειρήσεων, της σεξουαλικής κακομεταχείρισης και της βίας, καθώς και τις νέες γυναίκες οι οποίες έχουν ενσωματωθεί σε προγράμματα ενημέρωσης είναι κάτι το οποίο μπαίνει στην αρμοδιότητα των δικών μας προγραμμάτων. 10 εκατομμύρια ευρώ έχουν αφιερωθεί σε αυτά τα προγράμματα για την Τανζανία και την γύρω περιοχή. Η στρατηγική μας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η συνεργασία μας με άλλους ΜΚΟ και οργανισμούς οι οποίοι προστατεύουν τις νέες γυναίκες, τις νέες μητέρες, και η συνεργασία μας ε, με τα Ηνωμένα Έθνη και τα αντίστοιχα προγράμματα είναι κάτι που θα συνεχιστούν και το 2018. Ενσωματώσαμε τα προγράμματα αυτά όλες τις ε, νέες κοπέλες, ε, τις νέες μητέρες, νεαρές γυναίκες οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες των προστατευόμενων ατόμων. Το 2018 φυσικά και θα συνεχίσουμε τη δράση μας και θα ενσωματώσουμε και την αξιολόγηση των αποφάσεων της ε, κυβέρνησης της Τανζανίας για τις νεαρές ε, γυναίκες και τα νέα κορίτσια που γίνονται μητέρες στη Τανζανία. Είναι πολύ σημαντικό για μας να δούμε πώς εξελίσσονται τα θέματα των ε, παιδικών γάμων της ε, ίσης μεταχείρισης ε, ανδρών και γυναικών, κοριτσιών και αγοριών και ιδιαίτερα σε περιοχές της υπαίθρου έχουμε στηρίξει προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών για τις περιοχές αυτές και συνεργαζόμαστε με μη κυβερνητικού οργανισμούς θα ήθελα να σας πω ότι τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας έχουν ε, ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Είναι πολύ σαφής η απάντησή σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά τα προγράμματα φυσικά εξελίσσονται όπως μας είπατε. Παρόλα αυτά, Βλέπουμε ότι συνεχίζουν οι εγκυμοσύνες πολύ νέων ε, κοριτσιών και όλα αυτά θα έχουν επιπτώσεις ε, και στο άμεσο μέλλον. Τι ε, χρηματοδότηση προβλέπετε για τα επόμενα χρόνια σε αυτή τη χώρα. Έχουν οι νέες γυναίκες πρόσβαση στο οικογενειακό προγραμματισμό. Αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα το ποσοστό των κοριτσιών που είναι έγκυες και των κοριτσιών που είναι νέες μητέρες είναι τεράστιο. Και βεβαίως οι επιπτώσεις αυτών των, ε, αυτής της πολύ πρόορης εγκυμοσύνης είναι κάτι που φυσικά πρέπει να αξιολογηθεί για τα επόμενα χρόνια. Ναι, βεβαίως πρέπει και εμείς να δούμε, να μάθουμε, λέει η Πρόεδρος, και να επιλέξουμε ποια είναι η πιο σωστή προσέγγιση. Ευχαριστώ. Η Μαρία Χόιμπακ έχει κάνει επίσης μια ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που αφορά την συνάντηση με τα Ιδρύματα στις 19 Μαρτίου με διάφορα Ιδρύματα. Πρόκειται για φιλανθρωπικά ιδιωτικά ιδρύματα. Ποιος θα απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Μπέντο λέγομαι από την Μονάδα για την Κοινωνία των Πολιτών και τα σχετικά ιδρύματα. Ευχαριστούμε για την ερώτησή σας κυρία Χόιμπουχ και για το ενδιαφέρον σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των Ιδρυμάτων σε σχέση με την ανάπτυξη. Είναι καταλήτες καινοτομία, έρευνα, υπηρεσίες για δημοκρατία, για εκπαίδευση. Διάφορα μοντέλα έχουν αναδειχθεί. Πολιτικά, ιδρύματα, εταιρικά, κοινοτικά. Ε, ιδιωτικά για προώθηση των βιώσιμων στόχων, ψάχνουμε διάφορους τρόπους συνεργασίας, με αυτά τα ιδρύματα τα αναπτυξιακά, διάλογο, εταιρική σχέση, συνεργασία δηλαδή και με άλλους εμπλεκόμενους και οργανώνουμε την πρώτη συνάντηση. Να δούμε με τα κρατημέλη τι συνεργασία υπάρχει με τα ιδρύματα. Ανταλλαγή εμπειριών. Αυτό το, ήδη το κάναμε τέλη Ιανουαρίου. Και τώρα θα κάνουμε τη συνάντηση που αναφέρεται. Να δούμε τι τη θέμενη αξία θα υπάρξει. Και έτσι θα συνδυάσουμε δίκτυα διεθνή, σε εθνικό επίπεδο, Ευρώπη και σε περιοχές κόσμου στις οποίες εργαζόμαστε. Θα καλέσουμε και άλλους εμπλεκόμενους. UNDP, τον ΩΣΑ, μας βοηθήσουν με την εμπειρία τους. Να δούμε τι πνεύμα διαπνέει τη συνεργασία. Πώς να το να συνεχιστεί το έργο το οποίο ήδη έχει επιτελεστεί. Να δούμε σε τι άλλους τομείς μπορούμε να συνεργαστούμε και να δούμε τι συγκεκριμένα διαβήματα θα αναλάβουμε. Θέλουμε πιο στρατηγική προσέγγιση αυτών των εμπλεκομένων να ευθυγραμμιστεί η δράση απάντων όσον αφορά την υπόθεση, το μέτωπο της ανάπτυξης. Χόιμπουχ. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Αλλά δεν ξέρω για ποιες ε, συγκεκριμένες ε, προσκλήσεις ε, αναφέρεστε. Ποια ιδρύματα ακριβώς έχετε προσκαλέσει. Ποια ιδρύματα είναι ακριβώς αυτά που θα έρθουν. Ευχαριστούμε για την ερώτησή σας. Να, να σας πω, να σου ποια είναι τα ιδρύματα. Ε, αλλά εμείς δουλεύουμε μόνο με δίκτυα, γιατί θεωρούμε ότι έτσι η κοινωνία των πολιτών ε, εμπειρής αρμοδιότητας της μονάδας. Να σου πω, Worldwide Initiative, Wings, φιλανθρωπικό Charities, Community Foundations, Donors and Foundation Networks της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ιδρυμάτων, European Venture για Φιλανθρωπία και ο σχετικός φορέας, πολιτικά ιδρύματα,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 Grandmakers East Forum and then, as I've mentioned... Και επίσης το Ερμενέθρη με τον NDP και ο ΣΑ, όπως είπα στην αρχή. Μαρία, καλύπτωσε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, για την ενημέρωση. Και έτσι ολοκληρώνει τη των ερωτήσεων. Και πάμε τώρα στα διάφορα. Θα με 23 δεν μου είπατε για τίποτα για τα διάφορα. 27 Φεβρουαρίου. Έχουμε κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Γεωργίας όσον αφορά τις επιπτώσεις της ε, αναπτυσσόμενης χώρες της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής. Πρέπει να έρθετε σε εκείνη τη συνεδρίαση. Εγώ δεν μπορώ, αλλά όλοι οι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει θα πρέπει να είναι εκεί. Ένας τουλάχιστον από κάθε πολιτική ομάδα. 6 Μαρτίου. Πολύ σημαντική συνάντηση στις 8.30 το πρωί έκτακτη συνεδρίαση, συνάντηση με τον πίτροπο Μίμητσα όσον αφορά τον διαρθρωμένο διάλογο και κλεισμένων και κατόπιν 19 Μαρτίου. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση αλλά είμαστε εδώ από τις 2.30 ε, και ευχαριστούμε τους γερμήνες. Ε, σας. και κι εσείς ε, λίγη ώρα και όλοι οι υπόλοιποι.